Καλημέρα συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Στις 14 Οκτωβρίου ενέκρινε η Επιτροπή την τρίτη εφαρμοστική έκθεση και θα ακούσουμε την παρουσίαση Λίαν Συντόμος. Το 2018 συντάξαμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα εμπορικά. Η συγγήτρια ήταν η κυρία Σάιφη τότε και είχαμε γύρει κάποιες ανησυχίες για το σχετικά χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης των εμπορικών προτιμήσεων στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε και θέσει και κάποια ερωτήματα. Είχαμε γύρει κάποια σημεία δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εμπορική πολιτική σε ορισμένους τομείς. Φαίνεται σήμερα ότι το ποσοστό αξιοποίησης, ο ρυθμός αξιοποίησης έχει ενταθεί, έχει βελτιωθεί. Όμως, παλιά οι συζητήσει ήταν πολύ τεταμένες, ειδικά για τη ΣΕΤΑ. Συνεχίζει να είναι το ποσοστό αυτό στο 36 περίπου της 100. Παρά τις προσπάθειες, τις εργασίες, τη δουλειά που κάναμε για αυτή τη συμφωνία, δεν επαρκεί αυτό το ποσοστό. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Γεραλντίν Έμπεργκερ για να μας παρουσιάσει την ε, έκθεση υλοποίησης και να μας σχολιάσει αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθετε σήμερα για να παρακολουθήσετε την παρουσίασή μας. Πέρσι ήταν η δεύτερη χρονιά που κάναμε έκθεση, φέτος είναι η τρίτη ετήσια έκθεση που συντάσσουμε και που εγκρίνουμε, εγκρίθηκε περίπου πριν από τρεις εβδομάδες, με ένα πολύ εμπεριστατωμένο έγγραφο εργασίας. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να αυξήσει τη διαφάνεια και να αναφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώ λειτουργούν στην πράξη οι εμπορικές τη συμφωνίες. Και αυτό το πράττουμε μέσω των εκθέσεων που ανακοινώνουμε και δημοσιεύουμε. Το πράττουμε διότι θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά και γιατί θέλουμε να εξετάζουμε τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε και να το συζητούμε μαζί σας. Θα ήθελα πρώτα να πω δύο λόγια για το πεδίο που καλύπτει αυτή η έκθεση, ποια είναι τα νέα στοιχεία συγκριτικά με την περσινή αντίστοιχη, καθώς και για το ποια είναι τα κύρια ευρήματα ως προς τις εμπορικές ροές, την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας, το ποσοστό αξιοποίησης και να θίξω ορισμένου τομεί τους οποίους παρακολουθούμε εκ του στην Επιτροπή Ίντα και εσείς ε, και το Κοινοβούλιο τη γεωργία, το εναϊφόρο ανάπτυξη, τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις και τα εμπόδια στο εμπόριο. Είναι όλα αυτά τα θέματα που σας παρακολουθούν και τα, τα παρακολουθείτε και εσείς στενά. Αυτό το μοντέλο λοιπόν θα ακολουθήσει η παρουσίασή μου. Στην έκθεση δεν ασχολούμαστε με όλες τις συμφωνίες και τις 41 ε, που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολούμαστε με τις 35. Είναι οι βασικές προτιμησιακές συμφωνίες. Υπάρχουν και συμφωνίες μη προτιμησιακής φύσης και συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες δεν καλύπτονται στην έκθεση αυτή, δεν βρίσκονται. Εάν τη διαβάσετε, και όποιος ενδιαφέρεται μετά την παρουσίασή μου ευχαρίστω ε, να του δώσω ένα αντίγραφο εδώ αυτού του φυλαδίου γιατί μόλις τώρα το δημοσιεύσαμε. Έχουμε και περισσότερα άλλωστε στο γραφείο μου. Η δομή της έκθεσης και τα κεφάλαιά της είναι παρεμφερή, μοιάζουν πολύ με την περσινή, με αυτό που λάβατε πέρσι, για να έχουμε συνέχεια το κάνουμε αυτό. Βεβαίως δεν αποκλείουμε να αλλάξει αυτή η μορφή με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη θέση του Trade Enforcement Officer, ο οποίος θα έρθει εδώ του χρόνου για να κάνει αυτή την παρουσίαση και θα είναι ο δικός σας ομόλογος για την εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου. Τέσσερις είναι οι κατηγορίες συμφωνιών Έχουμε τις σύγχρονες συμφωνίες νέας γενιάς. Εκεί περιλαμβάνουμε τις ε, δασμολογικές προτιμήσεις και τα μη τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, αλλά και κανόνες για την παροχή των υπηρεσιών, για την ε, ε, απελευθέρωση, για τον ανταγωνισμό, για το εμπόριο και την αηφόρα ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Μετά έχουμε τις, συμβάσεις, τις συμφωνίες πρώτης γενιάς που συνήφθησαν πριν από το 2006 με προτιμησιακές συμφωνίες με τους πιο σημαντικούς εμπορικούς μας εταίρους. Η Ελβετία, για παράδειγμα, η Νορβηγία, η Τουρκία, όλα αυτά είναι με συμφωνίες πριν από το 2006. Έχουμε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, με τους γείτονές μας εξ Ανατολών και έχουμε και τις 31 προτιμησιακές συμφωνίες με τους 31 προτιμησιακούς εταίρους για τις χώρες ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού. Νομίζω ότι έχοντας ε, αναφερθεί στις ομοιότητες με την περσινή έκθεση είναι χρήσιμο να αναφερθώ τι επιπρόσθετο καλύπτουμε ε, φέτος. Έχουμε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος για την εφαρμογή της ΣΕΤΑ. Στην περσινή έκθεση είχαμε ένα μικρό υποκεφάλαιο που μιλούσαμε για την προετοιμασία για τη θέση σε ισχύ της ΣΕΤΑ. Αντίστοιχα έχουμε μεριμνήσει για να έχουμε ίδιο περιεχόμενο για την συμφωνία με την Ιαπωνία που άρχισε να ισχύει τον, 1η Φεβρουαρίου του 2019. Έχουμε ένα οριζόντιο τμήμα για τη γεωργία και την, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και έχουμε και κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη. Και έχουμε και ένα κεφάλαιο για την ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις βοηθήσει. Όπως είπατε και εσείς για την ε, προτιμησιακή αξιοποίηση των ποσοστών αυτών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, αντί για 20 έχουμε 26 εταίρους φέτος που έδωσαν δεδομένα που μας επέτρεψαν να υπολογίσουμε το ποσοστό για τις εξαγωγές και αυτό είναι, συγκαταλέγεται στα θετικά. Υπάρχει μια διαφορά, μια εξέλιξη που θα ήθελα να τονίσω. Το μερίδιο τις εμπορικές δραστηριότητες με τους προτιμησιακούς μας εταίρους ε, ε, βρίσκεται σε άνοδο. Έχουμε καλύψει περίπου το 31% του εξωτερικού εμπορίου με βάση ε, τις συμφωνίες μας με προτιμησιακούς εταίρους. Αν συμπεριλάβουμε και τη συμφωνία με την Ιαπωνία φτάνουμε στο 34% και αν επρόκειτο να συμπεριληφθούν εκεί και οι συμφωνίες με τη Μερκ Κοσούρ, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, αν καταφέρουμε, θα φτάσουμε στο 40%. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα κινούνται και όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτά το, η εμπορική δραστηριότητα που εκτελήσεται με βάση τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τους προτιμησιακούς μας εταίρους και γι' αυτό είναι κοινή ευθύνη των μελών και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να κάνουν όλοι το παν για να μπορέσουν να είναι λειτουργικές τέτοιου ίδιου συμφωνίας. Αυτό που επίσης ενδιαφέρει, το είπα και προηγουμένως, είναι το εξής. Έχουμε τους τρεις βασικούς εμπορικούς μας εταίρους. Η Ελβετία, για παράδειγμα, το 27%. Η Τουρκία και η Νορβηγία περίπου στο 11% είναι οι τρεις βασικοί μας εταίροι. Τώρα στις υπηρεσίες η Ελβετία καταλαμβάνει πολύ περισσότερο, 40% του προτιμησιακού εμπορίου, 9% η Νορβηγία, 7% ο Καναδάς, 6% η Τουρκία και 5% η Νότια Κορέα. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας εταίρη και το ίδιο περίπου ισχύει για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Πρώτον η Ελβετία, μετά η Τουρκία και μετά η Νορβηγία. Κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όπως και πέρσι το 2018 και φέτος ε, το εμπόριο με τους προτιμησιακούς μας εταίρους είναι σε άνοδο. Γενικά κατά 3,2% είχαμε αύξηση το 2019 και αύξηση εξαγωγών περίπου κατά 2% και εισαγωγών αύξηση κατά 4,6% περίπου. Αυτό ισχύει και για τα αγροδιατροφικά προϊόντα και για τα βιομηχανικά προϊόντα. Τα αγροδιατροφικά προϊόντα αυξήθηκε η εξαγωγή τους στις γειτονικές χώρες. Μιλούμε για συμφωνίες δεύτερης γενιάς, π.χ. με τον Καναδά συν 4%, με την Νότια Κορέα συν 4,8% και κυρίως και ιδιαιτέρως με τις γειτονικές μας χώρες εξαναλτολών συν 11% για Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία αλλά και τα βιομηχανικά ε, προϊόντα, εξορρυκτικά προϊόντα συν 20%, βασικά μέταλλα συν 4% και χημικά τρίτο στη λίστα εξαγώγημο αγαθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν 2,5% με βάση τις πρωτοημισιακές συμφωνίες. Ο, το μηχανολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε, τέλμη, σε τέλμα ως προς τις εξαγωγές και έχει μια πολύ μικρή υποχώρηση. Σήμερα, για πρώτη φορά, σε σχέση με φέτος είχαμε ένα ελαφρό εμπορικό έλλειμμα ε, της τάξης των 24,6 δις. Σε σύγκριση με αυτό, βάσει με, τις, με βάση τη ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου είχαμε πλεόνασμα 85 περίπου δις. Ε, μιλούσα για το εμπόριο και για τις εξαγωγές και για κάποιους από τους βασικούς εξαγωγικούς μας τομείς οι οποίοι είδαν την δραστηριότητά τους να αυξάνεται την τελευταία χρονιά αν και αυξήθηκε με πιο βραδύ πιο βραδύ ρυθμό από ότι το 2016-2017. Και εδώ θα ήθελα να σας δείξω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τους λόγους για αυτή την αξιολόγηση. Υπάρχουν κατασκευαστές οι οποίοι πράγματι συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας μας. Η κατάσταση έχει ως εξής. Το εμπόριο με τους προτιμησιακούς μας εταίρους αυξάνεται σε σχέση με το 2018 και θέλω να σας πω ότι εξετάσαμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία. Συνολικά το 2018 Το οικονομικό κλίμα ήταν τεταμένο, είχαμε τις κυρώσεις, είχαμε την κρίση του πολυμερού συστήματος, πάρα πολλά εργοτάξια και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Επιπρόσθετα, είδαμε κάποιους από τους βασικούς προτιμησιακούς μας εμπορικούς εταίρους και τις εξελίξεις που θα μπορούσαμε να έχουμε με αυτούς. Θέλω να ξεκινήσω με την Νότια Κορέα, η οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ε, το 50% των εξαγωγών μας με βάση τις συμφωνίες δεύτερης γενιάς κατευθύνεται στην Νότια Κορέα. Το 2017 είχαμε 30% εξαγωγές, ενώ φέτος μειώθηκαν οι εξαγωγές κατά 1% προς την Νότια Κορέα. Εξετάσαμε το θέμα και βρήκαμε κάποιους λόγους που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν. Ασθενή ζήτηση στην Νότια Κορέα. Η ζήτηση μειώθηκε κατά 9% υπερτίμηση του ευρώ σε σχέση με το κορεάτικο νόμισμα, αλλά και πολύ ισχυρό αποτέλεσμα βάσης. Δηλαδή το 2018 είχαμε τεράστια αύξηση εξαγωγών σε πολύ καθορισμένους τομείς ημιαγωγούς και αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων, ενώ την επόμενη χρονιά η κατάσταση ήταν σε τέλμα ή ε, σε μείωση, σε πτώση στους ίδιους κλάδους και μειώθηκαν οι εξαγωγές του μηχανολογικού εξοπλισμού, που είναι τα δύο βασικά εξαγώγημα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγχώρια ζήτηση λοιπόν μειώθηκε και αυτό οδηγεί σε μείωση των εξαγωγών κατά 1%. Εξετάσαμε επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο με βάση τις προτιμησιακές συμφωνίες που είναι η Τουρκία και εδώ υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτή την ασθενή μείωση. Υπάρχει το θέμα του νομίσματος. Υπάρχει η υποτίμηση της τουρκικής λίρας η οποία ήταν πολύ μεγάλη, 40% σε σχέση με το ευρώ συγκριτικά με πέρσι. Αλλά και άλλοι παράγοντες υπησέρχονται εκεί που έχουν να κάνουν με έναν αριθμό εμπορικών εμποδίων που έχει υψώσει η Τουρκία και που επηρεάζουν αρνητικά τις εισαγωγές στην Τουρκία ευρωπαϊκών εξαγωγικών αγαθών. Δεν υπάρχει ευθυγράμμιση με, τις, ε, με την τελωνιακή νομοθεσία, ειδικά ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αν δείτε κανεί την κατάσταση με την Τουρκία θα καταλάβετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη μαζί με τους εταίρους να, τα, να παρακολουθεί αυτά στενά. Και έχει ε, κάνει υποβάλει προσφυγή στον ΠΟΕ σε βάρος της Τουρκίας. Μιλούσα για τη σύγκριση μεταξύ 2018 και 2019. Θα ήθελα να δω τι συμβαίνει αν συγκρίνουμε τις προτιμησιακές συμφωνίες μεταξύ τους και πώς τις συγκρίνουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 2018 αναπτύχθηκε η εμπορική δραστηριότητα με τους προτιμησιακούς μας εταίρους κατά 3,2%. Λιγότερη ανάπτυξη σε σχέση με το 6,4% που αναπτύχθηκαν οι εμπορικές μας συναλλαγές με τους μη προτιμησιακούς μας εταίρους. Και αυτά τα στατιστικά στοιχεία επηρεάζονται ιδιαίτερως από το γεγονός ότι δύο βασικοί μας εταίροι εμπορικοί, οι οποίοι οι δυο μαζί εκπροσωπούν το 30% του ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες, ευθύνονται γι' αυτό και είχαμε ισχυρή αύξηση προς αυτές τις χώρες. Ας δούμε με λεπτομέρεια κάποιους από τους τομείς. Ε, έχουμε τον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος παραμένει από τους μεγάλους δικαιούχους των εμπορικών μας συμφωνιών. Οι αγροδιατροφικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 2,3% 5% με βάση τις συμφωνίες δεύτερης γενιάς, 11% με βάση τις συμφωνίες με τους γείτονές μας εξ Ανατολών στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους αγρότες μας να έχουμε αυτές τις συμφωνίες. Αν δείτε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, θα δείτε ότι οι εισαγωγές από τους εταίρους μας είναι κυρίως προϊόντα που είτε δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε δεν υπάρχουν, όπως π.χ. τα τροπικά φρούτα, ενώ τα ευπαθή προϊόντα δεν είναι ε, σε αγαθά που εισάγονται. αντίθετα, οι εξαγωγές είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Έχουμε ζωικά προϊόντα, κρέας, αυγά, 14%, ποτά, αλκοολούχα, πνευματόδη 13%, σιτηρά, 7%. Και έχουμε διάφορα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τρόφιμα ε, επεξεργασμένα και μεταποιημένα. Με βάση τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου θα ήθελα επίσης να τονίσω και κάποια άλλα στοιχεία. Θα μπορούσε κανείς ατέρμονα να μιλάει για το πόσο επωφελείς είναι αυτές οι συμφωνίες, όμως το 2018 έχουμε συν 4% εξαγωγές με βάση τη ΣΕΤΑ και είναι καλή η κατάσταση και με την Νότια Κορέα. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος κατά 12%. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλιο κρέας έχουμε σύν 20% εξαγωγές με όλους τους εταίρους μας. 16.000 τόνους, 2 τρίτα των συνολικών εξαγωγών. Είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός που πρέπει κανείς να θυμάται όταν μιλά για ευπαθή γεωργικά προϊόντα. Με την Αίγυπτο είχαμε 20% αύξηση στις εξαγωγές ζάχαρης λόγω της ε, κατάργησης του τέλους του δασμού των 20% σε αυτά τα προϊόντα. Μιλώ για τους δασμούς, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το IPR και για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων γεωγραφικές ονομασίες παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων και θα έλθω σε αυτά αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Με βάση τις σύγχρονες συμφωνίες μας με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, Συμφωνία με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, καλύπτονται διάφορα προϊόντα, 143 προϊόντα για παράδειγμα στη ΣΕΤΑ, στο, ε, στην εξυγχρονισμένη συμφωνία με το Μεξικό θα περιλαμβάνονται 340 προϊόντα. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να γίνουν είτε μέσω άμεσης προστασίας, είτε μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού που επιτρέπει στις εταιρείε να έχουν ξεχωριστούς μηχανισμούς εφαρμογής. Αυτά είναι τα δύο, αυτές είναι οι δύο διαδικασίες. Έρχομαι τώρα σε έναν άλλο τομέα τα εμπόδια στο εμπόριο, ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Βασικό πλεονέκτημα στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τους εταίρους του, να έχει διάλογο για πολύ συγκεκριμένα θέματα σε διάφορα επίπεδα και σε επίπεδο Υπουργείων και σε επίπεδο εμπορικών αξιωματούχων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και ειδικών για τα εμπόδια στο εμπόριο, είτε τα υφιστάμενα είτε αυτά που θα μπορούσε κάποιος να εγείρει. Το 2018 τονίζουμε λοιπόν διάφορους τομείς όπου σημειώνουμε πρόοδο και που έχουν καταργηθεί ορισμένα εμπόδια. Το τονίζουμε αυτό στην έκθεση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η Νότια Κορέα έχει άρει τους περιορισμούς της εισαγωγή βόλου κρέατος από τις κάτω χώρες και τη Δανία. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Η Χιλή άνοιξε την αγορά ε, κρέατος της σε περισσότερα κράτη-μέλη το Μεξικό κατήργησε πολλά, πολλή γραφειοκρατία για διάφορα οποροκυπευτικά μήλα και αχλάδια από την Ισπανία π.χ. Το Μεξικό περιέκοψε τον φόρο παροχής υπηρεσιών. Θα ήταν μεγάλο εμπόδιο αυτό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η Αίγυπτος ε, χαμηλώνει τους δασμούς σιγά σιγά για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και κατήργησε το τέλος και το δασμό για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και η Αίγυπτος ε, κατηρήσε και τους περιορισμούς στις εξαγωγές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Είναι λίγα παραδείγματα αυτά. Να θυμάστε όμως ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου παρουσιάζουν προκλήσεις και μπορούμε να σταθούμε στο ύψος και να απαλύνουμε, να μειώσουμε, να μετριάσουμε τα εμπόδια τα εμπορικά. Έχετε αναφερθεί στη ΣΕΤΑ και εσείς και εγώ θέλω να αναφερθώ στη ΣΕΤΑ. Ε, όλα τα διαχειριστικά εργαλεία εγκρίθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν το 2018. Οι περισσότερες επιτροπές πράγματι συνεδρίασαν το 2018. Και έχουμε τώρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής ε, εξελίσσονται οι ευρωπαϊκές εξαγωγές θετικά στο, ε, το εμπόριο αυξήθηκε κατά 10% γενικά. Αν δούμε όμως ορισμένους κλάδους που έχουν σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλάδοι που είχαν πολύ υψηλούς δασμούς πριν από τη ΣΕΤΑ, να δούμε τι έχει γίνει μετά την εφαρμογή της συμφωνίας οι εξαγωγές φαρμακευτικών αυξήθηκαν ε, κατά 13%, είναι το 12% των συνολικών μας εξαγωγών στο Καναδά και είχαν πολλούς δασμούς. Ε, τα αυτοκίνητα είναι το 11% των εξαγωγών μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Παρακολουθούμε κάποιους κλάδους όπου υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά η διαχείριση των ποσοστώσεων για βιομηχανικά αλλά και ε, παραδοσιακά ε, τυροκομικά προϊόντα. Και όντως δεν έχουμε διευκολύνει τους ε, ε, τυροκόμους να εξάγουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν ακόμα. Δεν ήθελα να αναφερθώ στο low preference utilization rate. Θα πρέπει όμως, γιατί το είπατε κι εσείς. Είδαμε τα στοιχεία του 2018 και είδαμε ότι αθρηστικά είμαστε περίπου στο 37%. Και αυτό είναι πράγματι χαμηλό. Αν συγκρίνουμε με άλλες συμφωνίες, με την Κορέα για παράδειγμα όπου το ποσοστό είναι κάπως υψηλότερο. Οφείλεται σε ένα αριθμό αιτιών, παραγόντων. Πρώτον, και σε γενικέ γραμμές. Να μην ξεχνάμε ότι το πρώτο έτος εφαρμογής, υλοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίες, μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα εκρεμή. Για παράδειγμα, με τον Καναδά, με τη ΣΕΤΑ, οι εταιρείε πρέπει να ετοιμαστούν να μπορούν να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες προέλευσης, στο νέο σύστημα τεχνολογίας και πληροφορικής. Μιλήσαμε με εταιρείε στην αυτοκινητοβιομηχανία, όλα αυτά τα δρομολογούν και τα κάνουν σιγά σιγά. Εξετάζουμε και την εξάλληψη της σταδιακή των δασμών για τα οχήματα. Είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δασμολογικού κύκλου. Οι εξαγωγές αυτοκινητών αυτοκινήτων αποτελούν το 14% όλων των επιλέξιμων εξαγωγών προς το Καναδά και αυτό έχει σημασία. Τώρα αν βγάλουμε τον τομέα των μεταφορών από τον υπολογισμό του ποσοστού τότε θα είχαμε ένα ποσοστό αξιοποίησης της προτιμησιακής αυτής συμφωνίας θα ήταν 40% ή και 55% φέτος. Δηλαδή ο τομέας των μεταφορών είναι που τραβάει το ποσοστό προς τα κάτω. Και στην έκθεση του αναφέρουμε ότι στη ΣΕΤΑ μπορεί κανείς αναδρομικά να ζητήσει αυτή την προτίμηση. Μπορεί ως εξαγωγέας, ως εισαγωγέας μάλλον στον Καναδά, έχει τρία χρόνια στη διάθεσή του να διεκδικήσει αυτή την ε, προτιμησιακή δασμολογική κατάταξη αναδρομικά. Είναι δύσκολο να γίνει δια, ε, ο διαχωρισμός μεταξύ αμυγός αγρο... αγροτικών προϊόντων και διατροφικών. Αλλά είναι λογικό τα γεωργικά προϊόντα να εισάγονται στο Καναδά με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ότι άλλα προϊόντα στην αρχή της εφαρμογής της οποιασδήποτε συμφωνίας. Θα ήθελα σε γενικές γραμμές να πω ότι η αξιοποίηση αυτού του πρωτοημισουιακού καθεστώτος, αν την εξετάζουμε αθρηστικά, αν τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι, δεν είναι αυτό καλός δείκτης για το πώς λειτουργεί η συμφωνία. Ε, γιατί υπάρχουν πολλές επιμέρους διαφορές που μας διαφεύγουν και αν θέλετε σας το αναπτύσσω αργότερα, αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Να πω για τη ΣΕΤΑ επίσης ότι δεν έχει σκοπό μόνο να εντείνει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, θέλει να προωθήσει τις ευρωπαϊκές αξίες και να λύσει παγκόσμια ζητήματα. Στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτέμβριο η, κοινή, Μικτή Επιτροπή οθέτησε τρεις συστάσεις για το εμπόριο και το κλίμα και τη Συμφωνία των Παρισίων για το φύλλο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τώρα ε, γίνεται μεγάλη συζήτηση μεταξύ των εταίρων για όλα αυτά τα θέματα και υπάρχει και ένα κανονιστικό φόρουμ κανονιστικών διατάξεων που ε, δημιουργήθηκε, που συνεδρίασαν τα μέλη του μία φορά και θα ξανασυνεδριάσουν στις αρχές του 20. Στα μέσα ε, Νοεμβρίου στην Οτάβα θα γίνει συνάντηση TST. Άρα η ΣΕΤΑ είναι μια συμφωνία που έχει σκοπό να προστατεύσει και να διαδώσει επίσης και τις αξίες μας. Ένας άλλος τομέας ή κλάδος που νομίζω θα σας ενδιαφέρει είναι το TSD, Εμπόριο και Φόρος Ανάπτυξη, που θα συνεδριάσουν τον Νοέμβριο και σε αρχές του 20. Επειδή έχω ξεπεράσει το χρόνο, το χρόνο που μου έχετε δώσει, θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ε, κάνουμε πολύ καλή πρόοδο Έχουμε ένα σχέδιο δράσης 15 σημείων ε, το 2018, τέσσερις βασικές προτεραιότητες των παραδοτέων. Δουλεύουμε σκληρά για να ενισχύσουμε τους διεθνείς ε, κανόνες για την εργασία, για το περιβάλλον. Αυτές οι δράσεις οδήγησαν στην κύρωση των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας από τρεις χώρες, Μεξικό, Βιετνάμ και Καναδά, για την ελευθερία του συνέρχεστε και του συνδικαλίζεστε και για τις συλλογικέ διαπραγματεύσει. Έχουμε κάποια παραδείγματα, Βιετνάμ, Ιαπωνία, ε, χώρες του Μερκοσούρ μεταξύ άλλων και βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες μας ουσιαστικά ενισχύουν το ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Δίνουμε στήριξη σε θέματα logistics, σε διάφορα έργα στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Έχουμε εγχώριες ομάδες συμβουλευτικής που σημειώνουν επιτυχίες. Στο Περού, για παράδειγμα, αλλά και στην Κολομβία, κυρίως στη Λατινική Αμερική, αλλά και στο Βιετνάμ. Δύο λόγια να πω για την επίλυση διαφορών και το EPA. Πέρσι, ορισμένοι ε, μου θέσατε ερωτήσεις για το EPA, για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και την επίδοσή τους. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη στις χώρες που είναι οι εταίροι μας. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των ε, συμφωνιών. Και υπάρχουν καλές εξελίξεις. Έχουμε 31 χώρες ΑΚΕ οι εξαγωγές τους σε εμά αυξήθηκαν κατά 5% στις 31 χώρες Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού. Είναι κάπως διαφοροποιημένες, όχι μόνο γεωργικά προϊόντα αλλά και προϊόντα μεταποίησης. 8% αύξηση στα προϊόντα τύπου ΝΑΜΑ. Όλο και περισσότερες χώρες συνάπτουν μαζί μας σε συμφωνίες εταιρικής και οικονομικής ε, σχέσης. Οι νήσοι αλλά και η νήσι Σαμόα, για παράδειγμα, είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και χρηματοδοτούμε διάφορα έργα και σχέδια για να διευκολύνουμε το εμπόριο μεταξύ χωρών και περιφερειών. Και ένα project είναι το, ε, μια διαδικασία διευκόλυνσης του εμπορίου στο Λεσότο, ε, στην πόλη Λεσότο, στην Αφρική, όπου είχαμε την ε, δημιουργία μιας απευθυντικής θηρίδας. Πέρυσι είχαμε μόνο μία παράγραφο για, την, ε, για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών και την επιβολή του νόμου. Ε, φέτος στην έκθεσή μας έχουμε περισσότερο περιεχόμενο στην έκθεση, ειδικά αναφορικά με την Κορέα, την Νότια Κορέα, την Ουκρανία, η οποία έχει μια απαγόρευση εξαγωγών που αντίκειται στην ε, Συμφωνία Σύνδεσης που έχουμε με την Ουκρανία και έχουμε και συμφωνία με την κοινό, αναπτυξιακή κοινότητα της Νοτιού Αφρικής. Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι περιορισμοί στις εξαγωγές πουλερικών οι οποίοι δεν δικαιολογούνται. Και έχει παραταθεί πέραν του λογικού ο περιορισμός αυτός που θα πρέπει να αρθεί. Ίσως να απαντήσω σε περισσότερα θέματα κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων και όχι μόνο στη βασική μου παρέμβαση και επίσης διάφορα άλλα θέματα έχουμε προσφυγές στο πλαίσιο του ΠΟΕ και όχι μόνο στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Συνοπτικά, οι προτιμησιακές συμφωνίες διευκολύνουν το εμπόριο. Ίσως χρειάζεται κάποιος χρόνος αρχικός να περάσει πριν φανεί αυτό. Είναι πολύ θετικοί παράγοντες ανοίγονται περαιτέρω διάβλη για επικοινωνία και για συζήτηση με τους εταίρους μας. Οι συμφωνίες αυτές μας επιτρέπουν να προστατεύουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, να συνεργαζόμαστε για κανονιστικά και ρυθμιστικά θέματα. Μας δίνουν τα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τις αντικσοότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμόρφωση και τέλος και εξίσου σημαντικό μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε και να καλλιεργήσουμε μια μακροχρόνια σχέση με τους εταίρους μας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλά εργαλεία, δεν δημιουργούν αυτόματα εκ του μηδενό εμπορική δραστηριότητα, αλλά είναι πολύ καλό που τα έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζω προσωπικά ότι ο διορισμός του Chief Trade Enforcement Officer θα βοηθήσει να αυξηθεί το κύρος, η δημοσιότητα, ε, η προσοχή που δίδεται σε όλη αυτή την υπόθεση, σε αυτό το φάκελο και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα και να επικοινωνούμε καλύτερα εμείς στην Επιτροπή με εσά στο Κοινοβούλιο. Και ελπίζω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να χτίσουμε μια ε, στέρεη εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους, την οποία θα αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω. Αυτά θα ήθελα να πω ε, προς το παρόν. Συγγνώμη που καθυστέρησα, δεν είχα καταλάβει ότι είχα λιγότερο χρόνο, νόμιζα ότι είχα περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, θα περιμένω για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Έχουμε ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αλλά και για την πολύ χρήσιμη γραπτή έκθεση για λόγους διαφάνειας όπως είπατε κυρία μου αλλά και για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή των συμφωνιών. Η σύναψη συμφωνιών όπως είπατε είναι κάτι θετικό για την οικονομία μας, για την πρόοδο των αξιών μας. Η παρακολούθηση όμως και η εφαρμογή είναι επίσης πάρα πολύ ε, σημαντικά στοιχεία και από αυτά που μας είπατε και διαβάσαμε φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δύο σχόλια για τη ΣΕΤΑ. Ποσοστό αξιοποίηση των ε, προτιμησιακών εξαγωγών ε, με τον Καναδά 37% μόνο. Θα ήθελα λοιπόν πιο συγκεκριμένα και πληρέστερα σε σχέση με την παρουσίασή σας να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι για το πολύ χαμηλό αυτό ποσοστό και νομίζω ότι ε, σαν κατακλείδα της παρέμβασής σας ε, κάνατε μια αναφορά στα μέτρα για την αύξηση αυτών των ποσοστών. Τι θα κάνετε, πώς θα πλαισιώσετε τις επιχειρήσεις, ε, πώς θα συνεργαστείτε περισσότερο με τα κράτη-μέλη, ώστε να πάμε λίγο πιο μακριά. Τα κράτη-μέλη είναι στην φάση της κύρωσης της ΕΤΑ, το υπενθυμίζω αυτό, άρα είναι καλή χρονική στιγμή. Δεύτερο, για τις δημόσιες ε, προμήθειες. Ε, ε, θεωρώ λυπηρό ότι δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για αυτά τα θέματα, και είπατε ότι υπάρχουν για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ΜΜΕ και πολλά άλλα θέματα, ξεχωριστά κεφάλαια. Το θέμα είναι σημαντικό για την Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε να προασπίσουμε τον βέλτιστο τρόπο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και για να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κριστόφ Χάνσεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή για αυτή την ε, ε, διεξοδική παρουσίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές ε, είναι περίπου το 86% των ε, επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβαίνουν σε εξαγωγές. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί δεν βλέπουμε το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των στοιχείων που παρουσιάσατε και ίσως μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα λεπτομερή στοιχεία μήπως δεν τα έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας πείτε ε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης η έκθεση πολύ σωστά επισημαίνει ότι το κόστος ε, ε, να μπει κανεί σε μία αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από από ό,τι για τις μεγάλες. Άρα δηλαδή ένα ε, μεγάλο εμπόδιο παραμένουν οι κανόνες ε, σχετικά με την προέλευση των προϊόντων. Άρα δηλαδή ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως προβλέπει κάποιο επιπρόσθετο εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί προέλευσης των προϊόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και το δικό μου το ερώτημα αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, που υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες και καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί περισσότερο το κεφάλαιο αυτό. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη μου αφορά στην καθοδήγηση ε, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξηγήσει διάφορα θέματα, προέλευση, δημόσιοι διαγωνισμοί, ε, πνευματικά δικαιώματα, όλα αυτά πολύ καλά, αλλά μήπως μπορείτε να κάνετε και κάτι για εκείνα τα θέματα όπου είναι πολύ πιο εύκολο για όλους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να προχωρήσουν. Ξέρω ότι είναι το θέμα ιδιαίτερα ε, περίπλοκο, αλλά ε, τι μπορείτε να κάνετε, όχι μόνο να περιορίζετε στην καθοδήγηση. Και το δεύτερο ερώτημά μου αφορά το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες συμφωνίες. Ε, βεβαίως είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό. Ε, ξέρω ότι με τη ΣΕΤΑ εκεί υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η συμφωνία για τις μικρομεσαίες, νομίζω κάπως έτσι αναφέρεται. Τέλος πάνω ένα κεφάλαιο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσθέθηκε μετά τη συμφωνία, αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία ΣΕΤΑ. Τώρα, σχετικά με άλλες ε, συμφωνίες, ε, μπορούμε να έχουμε ε, το θέμα των μικρομεσαίων επιχείρησεων να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή παρουσίαση και τα στοιχεία ε, πολύ ενδιαφέρον. Ε, και ήταν πολύ ωραίο να σας ακούμε να παρουσιάσετε την ομιλία σας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ασχοληθεί με το πώς μπορούμε να μετρήσουμε την πραγματική οικονομία. Το ΑΕΠ, ε, την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έχετε στοιχεία από αυτού και προτίθεστε να παρουσιάσετε στοιχεία τα επόμενα έτη. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά, με ενδιαφέρουν οικονομικές επιπτώσεις ε, σε αυτές τις συμφωνίες. Και μια δεύτερη ερώτηση, η Κομισιόν προβλέπει εξπόστα ε, μελέτη αντικτύπου σχετικά με τις ε, συμφωνίες αυτές, γιατί Ανησυχούμε πάρα πολύ για το ότι αυξάνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα μας ενδιέφερε ε, σε αυτές με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες πώς ακριβώς προκαλείται ενδεχομένω αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ενδελεχή μελέτη της. Ε, θέλω όμως παρόλα αυτά να ρωτήσω το εξής. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε μόνο στοιχεία ή μήπως πρέπει να αποδώσουμε περισσότερη σημασία στις πραγματικές επιπτώσεις που έχει το εμπόριο ε, στην γενικότερη οικονομική πολιτική κατάσταση μιας χώρας και γενικότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρθηκε ε, το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ελέγχθησαν. Αν δούμε όμως την πραγματικότητα στη Χιλή, στον Ισημερινό. Ε, και αν συγκρίνουμε αυτά, την πραγματική κατάσταση στις χώρες αυτές με αυτά που λέει η έκθεση, υπάρχει ένα χάσμα. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά που λέει η έκθεση και στην πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες. Τι συμβαίνει στους δρόμους. Άρα δηλαδή το εμπόριο οδηγεί στο να βελτιωθεί η κατάσταση ή μήπω ε, παροξύνει τι ε, διαφορέ και τι εντάσει ε, σε διάφορες χώρες. Ω εκ τούτου ενδεχομένως να πρέπει να εντάξουμε άλλα κριτήρια αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και ενδεχομένως να πρέπει να γίνει και μία συζήτηση, να μην ασχολούμεθα μόνο με το ΑΕΠ ως κριτήριο, και βεβαίω ε, για, να το, για να ε, ε, αξιολογήσουμε μέσω του ΑΕΠ και το εμπόριο, αλλά πρέπει το εμπόριο να το εντάσσουμε και σε μια ευρύτερη αξιολόγηση συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες. Εδώ εγώ ήθελα να κάνω απλά αυτή την γενικότερη παρατήρηση, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο τολμηροί, να εκμεταλλευόμαστε τις εκθέσεις με κάποια μεγαλύτερη τόλμη ε, και βεβαίως το θέμα της βιωσιμότητας ε, είναι <clears throat> καθοριστική σημασία ε, σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την ομιλία σας και επειδή έχουμε μια έκθεση από αυτού θα επανέλθουμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις περίπου προς μια κατεύθυνση που έκανε και ο κύριος Σόλτς. Ε, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για τις εισαγωγέ και τις εξαγωγέ, ε, που είναι πολύ ενδιαφέροντα, όμως εμά μας ενδιαφέρει το εμπόριο να έχει βιώσιμε επιπτώσει στις κοινωνίες μας και μία σημαντική ε, προέκταση του εμπορίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι σε ποια κρατημέλη, σε ποιες περιοχές προκύπτουν ε, ε, θετικές εξελίξεις λόγω εμπορίου. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι αυτά τα κεφάλαια ε, σχετικά σχετικά με τους στόχους χιλιετίας, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι και κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Έχουμε την πρώτη γενιά του κεφαλαίου, τα πρώτα κεφάλαια δηλαδή για το εμπόριο και την ανάπτυξη και έχουμε και τα πιο ε, εξελιγμένα, τα τελευταία. Εσείς βλέπετε να υπάρχει κάποια ποιοτική επίπτωση που να προέκυψε ειδικά από αυτά τα κεφάλαια. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω ε, πώς ακριβώς βλέπουμε την εκμετάλλευση μέσω του εμπορίου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω του, της νομοθεσίας κατά της δουλείας απαγορεύει στο σύνολό τους την εισαγωγή προϊόντων που έχουν παραχθεί με δουλική εργασία. Συγκεκριμένα παραδείγματα στη Μαλαισία. Εκεί υπάρχει ένα θέμα εξαναγκασμού εργασίας, δουλική εργασίας, ε, σε μια μεγάλη ε, μονάδα που παράγει ε, λαστιχένια γάντια για τα νοσοκομεία, αλλά και τα εξάγει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά στις Ηνωμένε Πολιτείε κανονικά δεν μπορούν να εξαχθούν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς τι, τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα του εξαναγκασμού σε δουλική εργασία. Η κυρία Χούπνερ. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω ανεπιφύλακτα ε, όλους τους αδέλφους που μίλησαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να προσθέσω και εγώ κάτι. Ε, όταν μιλάμε για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχει κάποια όθηση που να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως ε, και οι εταίροι μας έχουν κατανοήσει ότι είναι υποφελές ε, να λαμβάνουν ε, πιο σοβαρά υπόψη τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Ακούσαμε από εσά κυρίως στατιστικά δεδομένα. Εγώ δεν νομίζω ότι η έκθεση έχει ως στόχο μόνο το να παράγει δεδομένα. Είναι σημαντικό να γίνεται ανάλυση των στοιχείων και εγώ συμφωνώ με αυτό που που λέγεται ότι πρέπει να μπούμε πιο βαθιά, να προσπαθήσουμε να δούμε τις ε, προεκτάσεις των εμπορικών ανταλλαγών και για τις δύο πλευρές. Ε, όσον αφορά όμω τα στατιστικά δεδομένα, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί κάποια στιγμή συγκρίνατε το εμπόριο που βασίζεται στον ΠΟΕ με ε, με το εμπόριο που βασίζεται σε συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών και αν θυμάμαι καλά το πρώτο του ΠΟΕ μεγαλώνει και επεκτείνεται περισσότερο αυτό το εμπόριο από το άλλο. Η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, κατ' ουσίαν ε, ω το εμπόριο που τις αφορά στο σύνολό του αναλογεί στο υπόλοιπο εμπόριο που βασίζεται σε ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές. Εγώ σας ερωτώ, έχετε μια πιο βαθιά ανάλυση, πιο εντελεχή, πιο ουσιαστική. Γιατί το εμπόριο που βασίζεται σε, ελεύθερες, σε συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό που βασίζεται σε ρυθμίσεις του ΠΟΕ. Και μία άλλη ερώτηση. Όταν είπατε προηγουμένως ότι το 2018 ε, υπήρξε κάποια ανάπτυξη γιατί ήρθησαν ε, κάποιοι περιορισμοί. Αυτό δηλαδή ε, το ε, είπατε γιατί διαψεύσετε ότι συνέβη κάτι και μετά δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ πια ή μήπω διαφάνηκαν κάποιες μεσοπρόθεσμες τάσεις ε, ε, που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη και ενδεχομένως επειδή του χρόνου δεν θα, υπάρξουν, θα υπάρξει άρση άλλων εμποδίων, δεν θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Για μας είναι ενδιαφέρον να το ξέρουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τελευταία ερώτηση, αυτό στον Chief Enforcement Officer ε, αυτός ο αξιωματούχος, αυτή η θέση είναι επαρκώς ε, προετοιμασμένη, υπάρχει ήδη και τι μπορεί κανείς να πει σχετικά με το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπουρζουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την έκθεση και για την ανάλυση, για τα σχόλια ε, που ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα από τα στοιχεία. Ε, Όσον αφορά τις ε, γεωπολιτικές εξελίξεις, τον ε, προστατευτισμό, το άνοιγμα των αγορών, ε, το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες, το δικό μου το ερώτημα είναι, η εικόνα είναι ικανοποιητική, είναι αρκετά μεγάλη. Έχουμε δηλαδή αγορές όπου δεν υπάρχουν δασμολογικοί και εμπορικοί φραγμοί. Έχετε κάποια εικόνα για την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαστε ανταγωνιστικοί εναντί άλλων χωρών του κόσμου. Η, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότερες χώρες κατά μέσο όρο επενδύουν 2% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ε, ε, ανάπτυξη. Άλλες χώρες όμως επενδύουν μεγαλύτερο ποσοστό. Μήπως υπάρχουν λοιπόν εμπόδια ε, για τα προϊόντα μας που δεν είναι τελικά αρκετά ανταγωνιστικά. Έχετε έτσι κάποια άποψη από αυτού. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Τώρα το δεύτερο. Τα στοιχεία από τη Eurostat, εκεί τα στοιχεία ε, ανάμεσα σε στοιχεία για προϊόντα και στοιχεία για υπηρεσίες. Τώρα όμως βλέπουμε ότι το hardware και το software όλο και περισσότερο συνδυάζονται ε, συνδυάζονται όλο και περισσότερο τα προϊόντα με τις υπηρεσίες. Μεγατρόνικα. Έχετε εσείς ε, κάποια συγκεκριμένη άποψη σχετικά με αυτή την τελευταία εξέλιξη, τον συνδυασμό του hardware με το software. Και η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ, ε, κοιτάξτε, στην ε, παρουσίασή σας ε, κάνατε λόγο επανειλημμένα για κενά και υποτίθεται η λύση είναι αυτός ο αξιωματούχος, ο Chief Enforcement Officer, ε, σαν να είναι η μαγική αυτή λύση, αλλά εγώ ρωτώ η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή πότε προτίθεται να λύσει αυτό το μυστήριο. Ε, έχουμε 9 λεπτά στη διάθεσή μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε ακριβώς ε, στις 10. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω σε 9 λεπτά. Μεγάλη πρόκληση βέβαια να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά βεβαίω μπορούμε να συνεχίσουμε σε μικρότερο κύκλο αυτέ τι επαφέ. Για τη ΣΕΤΑ φυσικά και εξετάζουμε, τέλο πάντων εξετάσαμε τους λόγους, ήδη προανέφερα, ότι σε εξαγωγέ πρώτον άμα στον Καναδά έχουμε λάβει υπόψη μας ε, το μεταπητικό Χρειάζονται προσαρμογές για μεγάλους εξαγωγείς. Είμαστε σε επαφές με τις εταιρείες αυτές και κάνουμε ό,τι μπορούμε και από τις δύο πλευρές για να βελτιώσουμε την, ε, τα ποσοστά αξιοποίησης της ε, ΣΕΤΑ αλλά και των άλλων συμφωνιών. Δηλαδή, βελτιώνουμε το έργο μας ε, με δίκτυα τύπιος και υπάρχει και ένα εργαλείο που θα το καταθέσουμε σε αρχές του έτους για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά πρώτον ε, και θα έχουμε μία μοναπληθυντική πύλη. Δεν περιοριζόμαστε στις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών βέβαια. Θα υπάρχουν λοιπόν συνδέσεις σε εθνικούς ιστοτόπους ε, που είναι χρήσιμες πηγές και άλλες χρήσιμες πηγές. Για τις ΜΜΕ, πολλοί θέσατε ερωτήματα. Μεγάλη πρόκληση, το γνωρίζουμε. σε αδρές γραμμές για το 16 Ξέρουμε ποιο ήταν το μερίδιο των ε, ΜΜΕ που εξήγαν προς ε, τρίτες χώρες. 86% και 4% αξία. Δεν έχουμε στοιχεία για τα άλλα που είπατε. τα κεφάλαια ΜΜΕ δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη, είναι η απαρχή της συζήτησης. Μιλήστε για κάποιες συζητήσεις. Είπαμε στην Κοινή Επιτροπή ότι θα έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ορίσουμε επίσης συνδέσμους για τις ΜΜΕ στις δύο ε, διοικήσεις. Κάτι αντίστοιχο με το κεφάλαιο ΜΜΕ. Όλες οι νέες συμφωνίες περιλαμβάνουν κεφάλαιο ΜΜΕ. Ε. Με την Αυστραλία όπου να ολοκληρώνουμε το σχετικό κεφάλαιο. Άρα το γνωρίζουμε. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην έκθεση αναφέρω τη σχετική μελέτη για τις θέσεις που δημιούργησε το εμπόριο. Όχι μόνο οι προτιμησιακέ συμφωνία το 16. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. και δείχνει ότι από εξαγωγές εκτός Ένωσης εξαρτώνται 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μεταξύ του 2000 και του 2017 οι θέσεις που στηρίχθηκαν από όλες τις εξαγωγές, όχι μόνο δηλαδή τις προτιμησιακές, ε, ε αυξήθηκαν τα 66,1% ε, δηλαδή πάνω από 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Βέβαια, το είπατε κι εσείς, δεν είναι ε, τέλος στατιστικές, ε, είναι εκκίνηση πάνω στην οποία βασιζόμαστε. Όλοι μιλήσετε για τις στατιστικές όμως και ναι, ελπίζουμε να βελτιώσουμε τις αναλύσεις μας, να σας ε, εξηγήσουμε καλύτερα γιατί υπάρχει αύξηση ή μείωση εμπορίου. Βέβαια, ζητούμε την κατανόησή σας γιατί πολλά στοιχεία δεν σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή συμφωνών ελεύθερων συνάλλαγων, αλλά έχουν σχέση με άλλους παράγοντες. Θα δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα. Αλλαγή της ανταγωνιστικότητας με μερίδια σε ευρωπαϊκών τομέων, κλάδων στις τρίτες χώρες, έναντι άλλων τριτών χωρών ή οικονομικό περιβάλλον σε μια χώρα εταίρο. Για κάποιους εταίρους αυτό το κάνουμε ήδη. Συγκεκριμένα για την Κόρεα, την Νότια Κορέα. Το 18 είχαμε τη σχετική μελέτη ανάλυση των εξαγωγών και είχε και ένα κομμάτι για τις, εξαγω... για τις εκπομπές οξυδιού του άνθρακα. Για τις ε, ex post μελέτης αντικτύπου δεν μπορώ να σας απαντήσω. αλλά γίνεται για όλες τις συμφωνίες των αλλαγών πέντε χρόνια αφού τεθούν σε ισχύ. Για τα κεφάλαια εμπόριο βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε εξελίξεις, βλέπουμε ποιος είναι ο ποιοτικός αντίκτυπος. Υπάρχουν project τα οποία χρηματοδοτούνται για να υποστηριχθεί το έργο και κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η εκμετάλλευση των εργαζομένων τώρα. Όταν διαπραγματευόμαστε με τις χώρες, τους ζητούμε να επικυρώσουν τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας μεταξύ αυτών, τη Σύμβαση για την Αναγκαστική Εργασία. Δεσμεύονται όμως από τις βασικές αρχές ακόμη και αν δεν έχουν κυρώσει τις εν λόγω συμβάσεις. ΜΜΕ, πολύ ενδιαφέρον από του εμπορικού εταίρους, με τον Καναδά, παραδείγματο χάρη, Έχουμε επαφές για να δούμε πώς μπορούν οι ΜΜΕ καλύτερα να γνωρίσουν τα διάφορα εργαλεία. Στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη και υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον από τις ΜΜΕ. Για τη Eurostat νομίζω με ένα ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα όμως, ούτε και σε αυτό το ερώτημα. Θα δω τι σχέση υπάρχει μεταξύ λογισμικού και λογισμικού. Και το τελευταίο για τον Chief Enforcement Officer θα είναι το καθήκον της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόεδρος, Ursula von der στην ακρόασή της είπε κάποια πράγματα. Θα είναι ένας υψηλό επίπεδο αξιωματούχος, ε, που θα υπάγεται μάλλον στη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ εμπόριο και θα αναφέρει σε τίσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον Αρμόδιο Επίτροπο. Και ο ρόλος του θα είναι να ενισχύει ε, την εφαρμογή των εμπορικών δεσμεύσεων και των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών. Περιμένω και εγώ να δω ποιος θα πάρει αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αν ε, υπάρχουν συζητήματα που εκκρεμούν, δεν έχετε πάρει απαντήσεις, διμερώς μπορούμε να τα συζητήσουμε. Πρόεδρος, και να εμβαθύνουμε τη συζήτηση φαντάζομαι, γιατί σίγουρα ε, είναι στον αέρα ακόμη πολλά ερωτήματα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια ακόμη συνάντηση και συζήτηση για την υλοποίηση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Κλείνει εδώ η συζήτηση επί του σημείου 21. Και έχουμε το σημείο 22 που είναι η ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με μία μόνο ψηφοφορία για σήμερα. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, κάνω μία δοκιμαστική καταρχάς, ένα τεστ γιατί θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και πρέπει να έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. So, has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Είναι υπεράριθμο το ΕΛΚΑ ε, κατά έναν. Λοιπόν, πέρα τη δοκιμαστική ψηφοφορία. εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τώρα όμως θα περάσουμε στην πραγματική ψηφοφορία. Για τα πουλερικά. Στήθος Σκοτόπουλου από την Ουκρανία. Άρχεται ψηφοφορία. Ε, and... Okay, Πέρας. Εγκρίθηκε. ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 23. Δραστηριότητες των ομάδων παρακολούθησης. Οι ομάδες παρακολούθησης φυσικά και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Επιτροπής μας. Έχουμε 38 τέτοιες ομάδες παρακολούθησης. Και όπως είπα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Επιτροπής μας που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρουμε και πώς δουλεύουν, τι κάνουν και τι αποτελέσματα έχουν οι εργασίες τους. Έχουμε λοιπόν μονίμως αυτό το σημείο στη μέση διάταξη και το βάζουμε συνήθως μετά τις ψηφοφορίες ώστε να υπάρχει παρουσία πολλών συναδέλφων. Αλλά παρακαλώ για κάντε λίγη ησυχία. Όντα. Order που θα έλεγε και ο πρόεδρος του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, μετά τις ε, ψηφοφορίες συνήθως το βάζουμε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω για να είναι αρκετοί παρόντες και να ακούσουν τα περί των ομάδων παρακολούθησης. Έχουμε τέσσερις ομάδες παρακολούθησης που έχουν μέχρι στιγμής ε, συνεδριάσει. Η πρώτη αφορά την Ανατολική και την Νότια Αφρική. Χάιντι Χάουταλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes, ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, θα μιλήσω εκ μέρους της Έλξανς που είναι η μόνιμη εισηγήτρια και πρόεδρος της ομάδος παρακολούθησης για την Νότια και Ανατολική Αφρική. Έχω όμως ένα πρόβλημα. Μου έστειλε ένα μήνυμα αλλά δεν το βλέπω στην οθόνη μου ακόμα, οπότε δώστε με ένα λεπτό. Γιατί και εμείς ε, καταργούμε το χαρτί. Και στο Προεδρείο το καταργούμε, αλλά να, αφού δεν μπορώ, μου φέρανε ένα χαρτί. Είναι σαν ε, το παιδί του παπουτσί που δεν έχει παπούτσια. Λοιπόν, έγινε η πρώτη συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης για την ε, χώρες της Νοτιού και Ανατολικής ε, Αφρικής, στις 9 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Υπήρχε πλήρης εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων. Επίσης, υπήρχαν εκπρόσωποι της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο και ο πρόεδρος ε, της κοινοβουλευτικής ε, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Οι χώρες αυτές το Μαυρίκιο, με το Μαυρίκιο ε, αποφάσισαν να ξεκινήσουν ε, κάποιες συνομιλίες για την ενδιάμεση συμφωνία των συναλλαγών να είναι πιο εμβαθυμένη και να περιορίζεται στην πρόσβαση στην αγορά εμπορευμάτων. Θα υπάρχουν πιο ανατολικές ε, διατάξεις ε, για τις επενδύσεις, τις ενδείξεις, ε, τις δημόσιες συμβάσεις, τα πραγματικά δικαιώματα, τη γεωργία, το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρώτος γύρος συζητήσεων το Γενάρη και υπάρχει και ένας πολύ φιλόδοξος οδικός χάρτης με 45 γύρους διαπραγμάτευσης κατέτος και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ώστε οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2022. Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης λοιπόν, πολύ αποτελεσματική, ε, προβλήθηκε η σημασία της κλιματικής αλλαγής, ιδίω για τις νησιωτικές χώρες της ε, Ανατολικής Αφρικής, τονίστηκε η σημασία να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών, να λαμβάνονται υπόψη και να είμαστε και στο επίκεντρο όλων των διαπραγματεύσεων τα θέματα ισότητας των φύλων και οι εταίροι μας δεν θα πρέπει επίσης να γίνουν φορολογική παράδειση. Αυτό πρέπει να αποτραπεί. Επίσης ε, θα γίνει και μία μελέτη αντικτύπου ε, για τη βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι διαθέσιμα όμως πριν από δύο χρόνια. Στο μεταξύ θα συνεχιστεί η παρακολούθηση ε, της ε, αξιολόγησης αυτής. Είναι μια τερόκλητη περιοχή με ανισομερή ανάπτυξη. Η Έλλη περιμένει η επόμενη συνεδρίαση της μόνος παρακολούθησης για αυτές τις χώρες να λάβει χώρα. Έχετε ε, κοιτάξτε, ε, είχαμε μία συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου και το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ε, βεβαίως η απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τις ενισχύσεις που εδόθησαν για το Airbus και σχετικά με, τις, με τους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητήσαμε το όλο θέμα και αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι οι Ηνωμένες δεν δείχνουν καμία διάθεση να διαπραγματευτούν επί των δεσμών, διότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα και νομίζω Μάιο-Ιούνιο ε, θα έχουμε τη δική μας πρόταση σχετικά με τις ενισχύσεις ε, που έλαβε πέρυσι η Boeing. Ίσως λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και η λύση θα ήταν να έχουμε διαπραγματεύσεις, αλλά από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και νομίζω πολύ σύντομα θα έχουμε ε, άλλη μία ομάδα ελέγχου η οποία ε, θα εξετάσει το θέμα του ΠΟΕ και το θέμα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ε, δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τους ε, δασμούς. Γιατί αυτό το θέμα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική ομάδα παρακολούθησης. Δεν ξέρω, έχετε κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν έχετε ε, άλλες ερωτήσεις, πάμε στις Άζιαν, 15 Οκτωβρίου. Έχουμε εκεί την ομάδα παρακολούθησης. Λοιπόν, Πράγματι, η πρώτη συνάντηση τη ομάδα παρακολούθηση για τι χώρε ΑΖΕΑΝ ε, εστίασε την προσοχή τη στο κατά πόσο είναι δυνατόν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει με την Ταϊλάνδη. Όπω ξέρετε, ε, μεσολάβησαν οι εκλογέ και εμεί προσβλέπουμε σε μια πιο σταθερή κατάσταση ε, σε δημοκρατικέ εξελίξει. Πίτερ Μπέρτ, ο διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Trade, που ενεργεί, εκτελεί χρέη διευθυντή, ε, μας παρουσίασε την κατάσταση. Η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή αυτή και είναι η τέταρτη πιο πυκνοκατοικημένη στην περιοχή. Η οικονομία της ε, Ταϊλάνδης είναι διαφοροποιημένη, έχει ε, μεγάλη παρουσία η βαριά βιομηχανία και γίνονται και επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι η τρίτη σημαντικότερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ιαπωνία και την Κίνα. Βεβαίω πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολη αυτή η αγορά για τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζονται σε τοπικές δραστηριότητες γιατί ε, υπάρχει μεγάλη ευθερεσία που προβλέπεται από την νομοθεσία της ε, χώρας. Μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε το 2006 ε, συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών με τις χώρες της περιοχής. Το 2009 ελήφθη η απόφαση να διαπραγματευτούμε ξεχωριστές συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών με άλλες χώρες της περιοχής, ΑΖΕΑΝ, και αυτό το εξηγείται λόγω του ότι υπάρχουν και διαφορετικοί βαθμοί ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Οι διαπραγματεύσει με την Ταϊλάνδη μετά το πραξικόπημα του 2003 πάγωσαν και το 2017 είχαμε μια σταδιακή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με μικρές βελτιώσεις. Το Μάρτιο του 2019 είχαμε εκλογέ στην Ταϊλάνδη, συστήθηκε φέτο τον Ιούλιο μια νέα κυβέρνηση και ω εκ τούτου τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν τον Οκτώβρη προτείνουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αρκετά επιφυλακτική δηλαδή η όλη εξέλιξη. Και οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να δρομολογούν εσωτερικές διαδικασίες με διάφορους άμεσα ενδιαφερόμενους για να προετοιμάσουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούσαμε ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Άρα δηλαδή η Ταϊλάνδη πρέπει πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον η προτεραιότητά της είναι το TPP ή η ε, Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ταϊλάνδη πρέπει να σέβεται το, τη, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα θέματα της αλίας, γιατί εκεί ε, είχαμε μια εξέλιξη την άρση της κίτρινης κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2019. Πρέπει επίσης η Ταϊλάνδη να συμπεριλάβει άρθρα βιωσιμότητα τα οποία περιλαμβάνονται σε άλλε συμφωνίε ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών. Η όλη συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Οι βουλευτέ εξέφρασαν τι ανησυχίε του για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι εργασιακέ συνθήκε στη χώρα και σε κάποιε άλλε λεπτομέρειε τη συμφωνία και ένα θέμα το οποίο ετέθη ήταν η ε, χρήση της, ε, του εξαναγκασμού σε εργασία, κάτι το οποίο κάνουν ορισμένες εταιρείες στη χώρα. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της, γιατί κατ' ουσίαν ε, σημαίνει και εκμετάλλευση μεταναστών εργαζομένων. Και μάλιστα και πολλές φορές οι δικηγόροι των, και υπερασπιστές των μεταναστών εργαζομένων οδηγούνται σε δικαστήριο δικαστήρια, κάτι το οποίο είναι παντελώς απαράδεικτο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η εσωτερική διαδικασία στην Ταϊλάνδη. Η δική μας θέση βασίζεται στην εντολή του 2006 και στην εντολή για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αισιόδοξη σχετικά με τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων λόγω του ότι έχουμε την παρουσία και της Σιγκαπούρης και του Βιετνάμ παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ταϊλάνδη είναι πολύ πιο δύσκολη περίπτωση και θα χρειαστούν περίπου 3-4 χρόνια για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις. Για να ολοκληρώσουμε, Πιστεύουμε ότι η Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή προτιμά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αυτή με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν ερωτήσεις από αυτού και περνάμε τώρα στην τελευταία ε, παρουσίαση για σήμερα στον κύριο Ντάντι που θα μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κύριε Πρόεδρε, χτες είχαμε την πρώτη συνάντηση με την ομάδα παρακολούθησης. Ήταν πολύ ουσιαστική αυτή η εργασία και ήταν και η πρώτη περίπτωση κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στις διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο. Ε, η ΟΠΟΕ ενδιαφέρεται πάρα πολύ, ε, αλλά και όλοι οι μεγάλοι παίκτες ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ρωσία, ε, οι παίκτες όλοι αυτοί ε, δεν περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις, ούτε και η Ινδία και η Νότιος Αφρική. Η δουλειά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις αυτές ο στόχος είναι να αυξηθούν οι ροές ηλεκτρονικού εμπορίου ανά τον κόσμο και να μην υπάρχουν αδικαιολόγητα εμπόδια διασυνοριακά. Να βελτιωθούν οι εμπορικές ανταλλαγές, να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των ε, ε, καταναλωτών, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η συγκεκριμένη στόχη. Και επ' βέβαια προσθέθηκαν και άλλα δευτερεύοντα θέματα, επί των οποίων επίσης γίνονται διαπραγματεύσεις. Και όλα αυτά ε, ξεκίνησαν ε, ουσιαστικά η Αυστραλία είναι η χώρα η οποία καθοδηγεί όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή η Αυστραλία καθόρισε ένα πολύ έντονο χρονοδιάγραμμα Υπήρξε ε, μία, ένας τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων πριν από δύο εβδομάδες. Ακολουθεί ένας άλλος γύρος διαπραγματεύσεων κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Θα υπάρξει και μία συνάντηση σε επίπεδο ε, πρεσβευτών περίπου το Δεκέμβρη. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που συζητούνται. Βεβαίως και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά οράματα από πλευρά των άμεσα ενδιαφερόμενων. Η Κίνα, ας πούμε, προσπαθεί ε, μέσα από αυτό το εργαλείο να ε, προβάλλει το δικό της το ρόλο στην ψηφιακή τεχνολογία. Το ίδιο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Προσπαθούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο ο οποίο ε, θα εγγυάται κάποια θέση ισχύω. Ω εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι θα παρακολουθούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα παρακολούθησης είχε ως ε, καθήκον να εξετάσει έτσι το γενικότερο πλαίσιο της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Perfecto. Πολύ ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Εάν όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά στις ομάδες παρακολούθησης. Πάμε τώρα στο σημείο 54. Ε, της ε, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση μία ώρα. Παρουσίαση των συμπερασμάτων τη αποστολή τη Ένωση στο Μπαγκταντέ. Γίνεται ειδική παρακολούθηση λόγω των γεγονότων πριν από κάποια χρόνια. Μιλούμε για το Σύμφωνο Σταθερότητας Εμείς ε, ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παρακολουθούμε στενά τη κατάσταση και θέλουμε να βελτιωθεί ε, η κατάσταση των εργαζομένων στο τομέα της ε, κλωστοφαντουργίας της κατασκευής ε, και συγγραφής ρούχων στο Μπαγκλαντές. Πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς θα προχωρήσουμε. Και μπορεί τώρα να γίνει συζήτηση. Μετά την αποστολή. Τη αντιπροσωπεία της Επιτροπής στον Μπαγκλαντέ τον περασμένο μήνα. Θα έχουμε την έκθεση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή και μετά ο πρέσβης του Μπαγκλαντές θα μας πει τη δική του πλευρά. Και θα έχουμε και κάποιο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων και των σωματείων και συνδικάτων για να έχουμε πλήρη εικόνα. Uh, now start uh, with giving the floor to the Commission uh, for minutes. Λοιπόν, πέντε λεπτά ε, ο καθένας για να έχουμε μία ώρα σύνολο. Σας παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο, κάντε μια προσπάθεια. Η Μαντλέν παρακαλώ καταρχάς. Καλημέρα σας. Όχι Μαντλέν, αλλά Νίκος γιατί ο Νίκος είναι αυτός που πήγε στο Μπαγκλαντές και έχει πολλά πιο πολλά να μας πει παρακαλώ. Ο πρόεδρος φυσικά. Οι σημειώσει μου δεν είναι σωστές. Δεν είχα γράψει Νίκος, αλλά ευχαριστώ να σας ακούσουμε. Νίκος, σε ακούμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να, ζητήσουμε, να συζητήσουμε για αυτό το σύμφωνο. Είναι η πρώτη συζήτηση στη νέα Επιτροπή ΙΝΤΑ το βάζετε το θέμα στην ημερήσια διάταξη πολύ γρήγορα μετά τη σύστασή σα σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό δείχνει ότι σα ενδιαφέρει ιδιαίτερω και αυτό μα χαροποιεί. Σα ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σα, για το ενδιαφέρον σα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό μιλάω γρήγορα και γι' αυτό θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Πρώτον, να σα παρουσιάσω το πλαίσιο για τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση, για τι δεσμεύσει, για τι πληροφορίε τη αποστολή που έλαβε χώρα πριν από δυόμιση εβδομάδε και δύο λόγια για αυτό το σύμφωνο πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερική δράσης, για το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι σαφές αυτό που είπατε, Πρόεδρε, και αλήθεια. Το Μπαγκλαντές, το Μπαγκλαντές είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος αυτών των συμφωνιών εταιρική σχέσης. Τα δύο τρίτα δρέπει από τα ωφέλη στο σύνολο. Επομένως, το EPA έχει συμβάλει τα μάλλα στην οικονομική ανάπτυξη του Μπαγκλαντές. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, για να έχετε και μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους, 20 δις εξαγωγές 2 δις ευρώ από σε δασμούς που δεν συλλέγονται, δεν εισπράττονται. Το EBA έχει βοηθήσει τον Παγκλαντές να αυξάνεται σε, με θεαματικό τρόπο ο ρυθμος ανάπτυξης ανάπτυξη 6-7% ετησίως και έτσι έχει μειώσει την κατάσταση απόλυτη ένδυα και ε, ε, υπερβολική φτώχεια στον μπαγκλατε Δημιουργούνται κάποιε θέσει απασχόληση σιγά σιγά, ειδικά στον τομέα της ενδυμασίας, τη κατασκευή ρούχων. 4 εκατομμύρια θέσει απασχόληση έχουν δημιουργηθεί και οι περισσότερε κατά 60% καταλαμβάνονται από γυναίκε. Άρα, το EBA συμβάλλει τα μάλα στην ανάπτυξη του Μπαγκλατές και έχει φύγει το Μπαγκλαντές θεωρούμε ότι το 2024 θα φύγει από το καθεστώς LDC. Είναι απόφαση βέβαια των Ηνωμένων Αθηνών αυτό, το, του ΟΗΕ, αλλά μάλλον το 2024 ο ΟΗΕ θα βγάλει τον, τον Μπαγκλαντές από τη λίστα με τα απολύτως ενδεή κράτη. Τώρα, η ενισχυμένη δέσμευση ξεκίνησε το 2017, Enhanced Engagement. Παρόλο που είχαμε αυτή την πηξίδα, αυτό το σύμφωνο από το 2013 και παρόλο που έχει σημειωθεί πολύ καλή πρόοδο σε θέματα ασφάλειας και υγείας, Πολύ λιγότερη πρόοδος έχει σημειωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα. Ενισχυμένη δέσμευση λοιπόν, διότι με βάση το EPA έχουμε μια σειρά υποχρεώσεων στους δικαιούχους για να εκπληρούν βασικές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν την ενισχυμένη δέσμευση παράλληλα με το σύμφωνο και το EPA. Θέλω να θυμίσω στην Επιτροπή σας ότι η συνεδρίαση για το Compact τον Ιούνιο του 2013 εκεί οδήγησε στις επίσημες αρχές του Μπαγκλαντές να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση να ευθυγραμμίσουν πλήρως την εργατική τους νομοθεσία με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Είχαμε διάφορα καταγγελτήρια από τη Γενέβη για ε, της καταστρατηγήσεις. Άρα έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στην νομοθεσία με τροποποίηση του εργατικού κώδικα στον Μπαγκλαντές από το 2018 μέχρι και την άνοιξη του 2019 που πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά σαφέστατα δεν αρκούν για να λύσουν όλα τα ζητήματα που έχει εντοπίσει ως πολύ προβληματικά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Αυτό ήταν το πλαίσιο λοιπόν της αποστολής μας που έγινε πριν από δυόμιση εβδομάδες, μια κοινή ε, αποστολή από πλευράς Επιτροπής και Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μαζί με το Τμήμα για την Απασχόληση και έχω και τον προϊστάμενο από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Και έγινε back to back με τις υποομάδες για το εμπόριο, για τη διακυβέρνηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανάπτυξη και για την εμικτή Επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκλαντές. Το γεγονός ότι επιλέξαμε και διαλέξαμε να έχουμε αυτή την αποστολή με αυτές τις συσκέψεις και συνεδριάσεις ήταν για να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ η πίεση στην κυβέρνηση. Και ε, νομίζουμε ότι καταφέραμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους βασικούς εταίρους, με τα συνδικάτα, με τα σωματεία, με τους εργοδότες, εκπροσώπους των εργοδοτών, με τις ΜΚΟ για θέματα εργασιακά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εκπροσώπους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών σημάτων, με τις ε, επιχειρήσεις του Μπαγκλαντές, BKMAIK, ε, με τη UNICEF, με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με εκπρόσωπο του ΦΑΟ, ε, και άλλου προσώπους διεθνών, οργανισμών. Είχαμε πολύ καλε συζητήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εμπορίου, Εργασίας, δικαιοσύνη και είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε με συμβούλου του Πρωθυπουργού. Είχαμε καλές συναντήσεις και σε όλες αυτές τις σκέψεις στείλαμε το μήνυμα ότι πρέπει τον Μπαγκλαντές να σημειώσει πρόοδο και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά δικαιώματα όπως καθορίζονται και όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Οργάνωση εργασία στις αντίστοιχε συμβάσει του. Τα καλά νέα. Είχαμε συμφωνία για τα επόμενα βήματα για τις συστάσεις και θα μιλήσω για τις συστάσεις για τα εργασιακά. Έχουμε ανάγκη να υπάρχει πρόοδος για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε, ε, να διαμορφώνονται σε εξαγωγικές ζώνες, ε, ειδικά αυτά στις εξαγωγικές ζώνες, στις ζώνες μεταποίησης ε, προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή άμεσα και να λυθεί και το θέμα της παρενόχλησης, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την παιδική εργασία. 1,2 εκατομμύρια παιδιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνεχίζουν να εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες στην άτυπη οικονομία, αλλά και αυτό θα πρέπει να λυθεί ω θέμα. Δεν θέλουμε μόνο το Μαγκλαντέ να ασχοληθεί με την επίσημη οικονομία. Και ω προ την επιθεώρηση εργασία, οι επιθεωρητέ εργασία. Η επιθεώρηση τη εργασία είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο γιατί χωρί σωστή επιθεώρηση δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σύμφωνοι ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται σεβαστά και τηρούνται. Τα καλά νέα είναι δηλαδή ότι έχουμε συμφωνία και οδικό χάρτη. Έχουμε συμφωνία να έχουμε οδικό χάρτη με τις βασικές αλλαγές με χρονοδιαγράμματα. Και αυτό είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας της επίπτωσης που θα έχουμε, το οποίο ανεφέρθηκε προηγουμένως. Και έχουμε και κοινή δήλωση μετά από την συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπαγκλατές. Όλα αυτά είναι επίσημα και δημόσια. Οι επιρρογνώμονες και οι δικοί μας θα συνεδριάσουν σύντομα για να δουν την εφαρμογή και την τήρηση του οδικού χάρτη. Ως προς το σύμφωνο τώρα, δεν συζητήθηκε αυτό αυτό στην αποστολή. Είναι παράλληλες οι διαδικασίες, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό άλληλο επικαλύπτονται. Τα καλά νέα είναι ότι παρατάθηκε η σύμβαση αυτή, η συμφωνία, μέχρι τα 2000 της επόμενης χρονιάς. Ήταν με τους κατασκευαστές BGMA και BKMA, οι βασικές επιχειρήσεις του Μπαγκλαντές, ιδιωτικέ ιδιωτικές στον τομέα της ενδυμασίας και της μεταποίησης και ε, ρούχων. Τώρα για το compact, για το σύμφωνο αυτό, ελπίζουμε το, η επόμενη συνάντηση να γίνει στην ΤΑΚΑ, την πρωτεύουσα, το πρώτο εξάμεινο του 2020 και συζητούμε τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Πώς θα διαβεβαιώσουμε ότι αυτές οι, πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι συνεδριάσεις είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι στο παρελθόν. Με αυτή τη σύντομη ε, δήλωση σταματώ εδώ για να μιλήσει και ο συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οχτώ λεπτά πήρατε εσείς, δύο λεπτά θα έχει ο συνάδελφός σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Το Μπαγκλαντές είναι ένα σημαντικός εταίρος στην περιοχή. Έχουμε διάφορες προτεραιότητες ε, τις οποίες προωθούμε με τον Μπαγκλαντές, περιφερειακή σταθερότητα, ανάπτυξη, άτυπη μετανάστευση, ε, καταπολέμηση της κρίσης των προσφύγων, της προσφυγικής κρίσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασική προτεραιότητα για, το για και τον Μπαγκλαντές και γι' αυτό επιμείναμε να έχουμε επιπρόσθετη συνεδρίαση της υποομάδας για την καλή διαχείριση και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αποκινούμε την υποομάδα για τις εμπορικές ανταλλαγές με βάση το Everything But Arms, οτιδήποτε εκτός από τα όπλα, ε, μεταξύ άλλων. Η αποστολή EBA και η υποομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σωστή διακυβέρνηση έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα σε πολλές ε, συζητήσεις υψηλού επίπεδου εκφράσαμε ξεκάθαρα τις ανησυχίες μας σε σχέση με τις εκλογές, την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, τις εξαφανίσεις, ε, τις δολοφονίες, τα βασανιστήρια, ε, τις εξαναγκαστικούς, καταναγκαστικούς γάμους, την παιδική εργασία, τη θενατική ποινή μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεσμεύεται να ευθετήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων από την Οικουμενική Καθολική Περιοδική Αναθεώρηση. Ε, συμφωνήσαμε να έχουμε ε, μετά την έκθεση των ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την, για τις εκλογές, ε, παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας. και στηριζόμαστε στη δέσμευση που έχει αναλάβει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πράγματι να ε, λειτουργήσει επικοδομητικά και να προωθήσει αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Um, Ωραία. Τώρα. Και εσείς μπορείτε να πάρετε το λόγο MSA για 5-6 λεπτά. Uh, thank you very much for Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Μπαγκλαντέ τα τελευταία χρόνια έχει ω αποτέλεσμα πολλές ε, επιτυχίες. Και τις προβάλλουν και τα διεθνή μέτια και εμείς. Είμαστε από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας η χώρα με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και σε ό,τι αφορά κοινωνικούς δείκτες, όπως ε, την χειραφέτηση των γυναικών, σε πολύ καλή θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει και σε υψηλό επίπεδο. Η Ροχίνγκια. Είχαμε την ανθρωπιστική κρίση της κοινότητας αυτής. Πάνω από το 62% ε, της, ε, των εξαγωγών είναι στην Ένωση. Ουσιαστικά είμαστε σαν ανάδοχο παιδί αυτού του μηχανισμού. σε σχέση με την παραδοσιακή βοήθεια που παρεχόταν από την Ένωση και έτσι πολλά εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας μας βγήκαν από το καθεστώς της φτώχεια. Πρέπει να τονίζουμε και τα ωφέλη αυτής της ε, συμφωνίας γιατί θα βοηθήσουμε να μην ε, προβληθούν κάποια προσχήματα ε, ότι οι δικαιούχοι της χώρες δεν κάνουν αυτό πρέπει. Οι πολιτικές τώρα. Βλέπουμε εξελίξεις στην κλωστεφαντουργία, αύξηση του κατώτατου μισθού, 162% είναι η αύξηση αυτή από το 2010 μέχρι σήμερα. καταγράφησαν 693 νέα συνδικάτα από το 2013 και μετά και έχουμε και 3.800 εργοστάσια που ε, τα επιθεωρήσαμε για να δούμε τις πυροσβεστικές ε, δομές για την ασφάλεια, την επαγγελματική και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν θετικά τα αποτελέσματα, πάνω από το 90%. Υπάρχει ε, υποχρεωτική Επιτροπή Επιθεώρησης της Ασφάλειας σε κάθε εργοστάσιο. Υπάρχει το μνημόνιο συνεννόησης για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στο ανεξάρτητο καθεστώς παρακολούθησης στην συγκεκριμένη βιομηχανία. Και έχουμε και το Συμβούλιο Βιωσιμότητας. now has world... Το Μπαγκλαντές πλέον έχει το μεγαλύτερο αριθμό πράσινων εργοστασίων. Και έχει πάρει και 25, έχει σε 25 περιπτώσεις έχουμε platinum κατηγορία. Και έχουμε αυξήσει το μερίδιό μας στην αγορά από το 2014 το 2018. Η πρόθεση της βιωσιμότητας ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος παραγωγής, το περιβαλλοντικό κόστος όμως ταυτόχρονα. Θα θέλαμε η υπεύθυνη πολιτική της Ένωσης να φροντίσουν, να μελετήσουν τα σχετικά, γιατί θέλουμε δίκαιες τιμές, σωστές τιμές, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα μόνο στην αγορά. Είναι προς όφελός μας, πιστεύω, και προς το συμφέρον μας να προωθήσουμε εξωπρεπή εργασία και ε, καλές εργασιακές σχέσεις στον τομέα της λουστεφαντουργίας στη χώρα μας. Έγιναν σημαντικές τροποποίησεις με τριμερείς διαβουλεύσεις και είχαμε και τον ε, νόμο των εργασιακό νωρίτερα φέτος. Έχουμε επίσης ε, συστάσεις από τον ε, εποπτικό μηχανισμό εργασίας, τις λαμβάνουμε υπόψη, το σύμφωνο βιωσιμότητα πρόσφατα συμφώνησε να προχωρήσει με οργανωμένο τρόπο στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης με τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς θα συμμετέχουν. Γι' αυτό και εξεπλάγημεν που κάποιοι εκπρόσωποι στο ΔΟΕ κατέθεσαν τον Ιούνιο καταγγελία χωρίς να έχουν ε, πρώτα έρθει σε επαφή με τους τοπικούς ομολόγους τους ε, στο Μπαγκλαντές. Πρόκειται για καταγγελίες οι οποίες έβρεθαν ανακριβιών και ψευδών πληροφοριών. Νομίζω τώρα 26 της ε, σύμβασης του ΔΟΕ μίλησαν για ένα forum shopping και εμείς θεωρούμε ότι Ναι, η Ένωση πρέπει να λάβει γνώση και να σημειώσει αυτές τις καταγγελίες, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβει υπόψη... Όχι, δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Ε, και αυτά που λέει η κυβέρνηση και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ή να εστιάσει στην ε, πλατφόρμα αυτή το σύμφωνο βιωσιμότητας ή να ενδιαφερθεί να ε, ρωτήσει και άλλους φορείς. Υπάρχουν παρόμοιοι μηχανισμοί και για τον Παγκλατές και για τη Μιανμάρ και αυτό μας πληγώνει. Γιατί η Μιανμάρ ε, έχει κατηγορηθεί για αμέλεια. At a time when συγγνώμη, έχει κατηγορηθεί για εθνοκάθαρση και γενοκτονία από τον ΟΗΕ. Και μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι με αυτούς. Και βέβαια θα περάσουμε από τις ελάχιστα τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες τις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες αδυναμίες, κάποια τροτά σημεία εν γενή στη χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε την, ε, το καθεστώς ε, GSP+, Plus, για να μην μειωθεί και η πρόοδος που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Ίσως τα κριτήρια εισαγωγής θα έπρεπε να ε, επαναπροσδιοριστούν στο πλαίσιο του GSP+. Ε, ολοκληρώνοντας, ε, σας καλώ όλους να επισκεφτείτε το Μπαγκλαντές για να δείτε από μόνοι σας, με τα ίδια σας τα μάτια, όλα αυτά που προσπάθησα στο λίγο χρόνο που είχα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος εισηγητής επίσης για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε. Ε, Εμεί εκπροσωπούμε τους ε, εισαγωγείς, ε, το λιανικό εμπόριο, ε, όσους καταναλώνουν κυρίως έτοιμα ρούχα, ηματισμό. Έχουμε περίπου 2.400 μέλη ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Και παρότι εισάγουμε αυτά τα προϊόντα και ε, εκμεταλλευόμεθα τις, ε, τους προτιμησιακούς δασμούς που ισχύουν για χώρες όπως με το Μπαγκλαντές, παρόλα αυτά προσπαθούμε να έχουμε ένα ανοιχτό εμπόριο, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους της χιλιετίας των ΗΕ. Κυρίως στο Μπαγκλαντές έχουμε ένα πρόγραμμα για τη χειραφέτηση των γυναικών ε, και αυτό ε, μας απασχολεί πολύ. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία, εκείνο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Μπαγκλαντές. Έχουμε ένα μέλος στην Steering Committee και περίπου το 50% είναι ξένα μέλη. Έχουμε λοιπόν διαπιστώσει ε, πολλές ε, βελτιώσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις ε, περί ασφάλειας από πυρκαγιές και άλλα θέματα ασφάλεια ε, στο Μπαγκλαντές. Τον Ιούνιο του 2020 τελειώνει, ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν και εμεί θα αποδώσουμε ιδιαίτερη ε, συμφωνία στην, ε, αντικατάσταση αυτής της συμφωνίας. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτή τη συμφωνία ελπίζουν να συνεχιστεί η ίδια κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να υπάρξει συνέχεια Ακριβώ λόγω του ότι η συμφωνία αυτή ήταν πολύ επιτυχημένη. Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν κάποια θέματα που μας απασχολούν, ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη εξουσία. Αυτό λοιπόν μας ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί το Συμβούλιο έχει έξι μέλη από την BGMBA, έξι μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέσσερα ντόπια, δύο από άλλες χώρες και έξι μέλη από τη Συμφωνία και προσβλέπουμε στο να είναι και μια ουδέτερη θέση ε, κυρίως ε, από την BILO. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρότι εμείς ε, διαδραματίζουμε συμπληρωματικό ρόλο όσον αφορά το της ασφάλειας στο Μπαγκλαντές. Παρόλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται χρήση της τεχνογνωσίας που υπάρχει για θέματα ασφάλειας, να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί και να βασιστεί στην τεχνογνωσία που έχει προκύψει λόγω της συμφωνίας υπάρχει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία ε, κάνει ανεξάρτητους ελέγχους σε όλα τα εργοστάσια ε, που είναι μέλη μας. Καλύπτουμε πάνω από 30 τομείς. Ασχολούμεθα με τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις, την δίκαιη αποζημίωση των εργαζομένων, ασχολούμεθα όμως και με την ασφάλεια. Και αυτή η ασφάλεια αφορά κυρίως ε, τα, κτίρια και τα θέματα των ε, πυρκαγιών. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση κατά τα τελευταία έτη όσον αφορά πυρκαγιές σε κτίρια. Ε, παλαιότερα μόνο το 23% των εργοστασίων στο Μπαγκλαντές επιθεωρούντο για θέματα ασφάλειας, ενώ σήμερα μιλάμε για πάνω από το 65% εργοστάσια στα οποία γίνονται επιθεωρήσεις άρα δηλαδή σημαντική βελτίωση. Όσον αφορά τώρα την ε, συμφωνία EBA, αυτή είναι πολύ σημαντική για μας, ε, γιατί ε, καταβάλλεται κάποια συνεισφορά. Παρότι βέβαια μας ανησυχούν κάποια ευρήματα της Επιτροπής, πρέπει να πω ότι δεν εκπλησόμεθα ιδιαίτερα. Στον Μπαγκλαντές διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο και παρότι έχουμε διαπιστώσει σημαντική βελτίωση σε θέματα ασφάλειας, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτά τα και να επιβάλλει το συντομότερο δυνατόν τις απαραίτητες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα ταχύτατα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι φέτος ξεκίνησε μία έρευνα ε, κατά της Καμπότζης. Τα αποτελέσματα θα τα ε, δείτε πολύ σύντομα και φοβάμαι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα δεν θα είναι ιδιαίτερα θετικά για την Καμπότζη. Τώρα, κατά πόσο θα ξεκινήσει περιττέρω έρευνα σε σχέση με την Καμπότζη, αυτό θα το αποφασίσει το ίδιο το Μπαγκλαντές. Εμείς ε, προτιμούμε να διατηρηθούν οι προτιμήσεις, γιατί αυτό ωφελεί τα μέλη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει αν η έρευνα καταδείξει και καταλήξει διαφορετικά συμπεράσματα, εμείς θα τα δεχτούμε, διότι η ο κώδικας ε, διοντολογίας, ε, τον οποίο δέχονται όλα τα μέλη μας, είναι άρρηκτα συνδεμένος με τις ε, διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νιούμαν και από πλευράς συνδικάτων έχουμε την κυρία Σαντ Σαχάν. Εμείς εκπροσωπούμε 270 εκατομμύρια εργαζόμενους. Έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις σχετικά με το τι ακριβώς διαδραματίζεται στον Μπαγκλατές τα τελευταία χρόνια. Είναι μία από τις δέκα χειρότερες χώρες του κόσμου για την παραβίαση της ελευθερίας του συνέρχεστε με βάση τις έρευνες που γίνεται κάθε χρόνο. Ε, υπάρχει επιδείνωση του δημοκρατικού χώρου για τους εργαζόμενους για να μπορούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη ε, δικαιώματά τους. Ε, τον ε, περασμένο Σεπτέμβρη ορίστηκε ένας κατώτατος μισθός, αλλά αυτός που δεν είναι δεν αρκεί για τους εργαζόμενους για να μπορούν να επιζήσουν. Η κυβέρνηση ε, όμως μοιάζει να αρκείται στο ότι θα υπάρχουν αυτοί οι μισθοί ε, της πείνας. Οι μισθοί καταρακώνονται. Είχαμε και φέτος ένα θάνατο και πολλούς τραυματισμένους ε, από συγκρούσεις ε, ε, πολλοί εκπρόσωποι εργαζομένων ε, έχουν δεχτεί αντίπεινα τουλάχιστον 52 ε, συμπεριλαμβανομένων και συνδικαλιστών συνελήφθησαν. Και αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα από την εφετινή χρονιά. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έχουν το δικαίωμα του συνέρχεστε για να μπορούν και να ζητήσουν, να διεκδικήσουν βελτίωση ε, των εργασιακών συνθήκων. Όσον αφορά την ασφάλεια, δεν υπάρχει πρόοδος. Η κυβέρνηση δεν έχει πράξει τίποτα για να βελτιώσει την ε, κατάσταση της ασφάλειας, κυρίως από πυρκαγιές. Τον Ιούνιο του επόμενου έτους ε, εκπνέει και σχετική συμφωνία. Επιπλέον, ε, ίσως να υπάρχει μία μείωση του αριθμού των θανάτων, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που υφίστανται τραυματισμούς ε, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν προσφέρει καμία ασφάλεια από τέτοιου είδους ατυχήματα. Το Μπαγκλατές εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερα ε, περιοριστικές ε, εργασιακές διατάξεις. Οι τελευταίες αλλαγές ε, στη νομοθεσία περιεργασίας δεν κάλυψαν τις ανησυχίες που υπάρχουν κυρίως σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεστε. Οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας κατέστησαν σαφές ότι θα συνεχίσουν να εκφράζουν αυτές τις επιφυλάξεις τους από 30 σε 20% έχει αυξηθεί μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων που είναι απαραίτητος ε, για να μπορεί να συσταθεί με ένα εργοστάσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο και αυτό ανησυχεί κυρίως ε, όσον αφορά τις ε, καταστολές, βίες καταστολές σε διαμαρτυρίες για ε, μισολογικά ε, αιτήματα και μισολογικές διεκδίκεις. Um, σε ζώνες όπου γίνονται εξαγωγές οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην μπορούν να συστήσουν συνδικάτα και οι επιτροπές εργασίας δεν μπορούν να επισκεφτούν τα εργοστάσια χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αναγγελία. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια παραμένουν απαράδεκτα. Βεβαίως όλα αυτά δεν είναι άγνωστα στην κυβέρνηση, τις, ε, τα έχουμε επισημάνει, ε, τα έχουν επισημάνει και όλοι οι εκπρόσωποι του ΔΟΕ, αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος τα τελευταία δέκα χρόνια και όπως είπε και ο πρέσβης, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΛΟ έχει καταθέσει διαμαρτυρία εναντί του Μπαγκλαντές γιατί παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και έχει συστήσει μία ε, ερευνητική επιτροπή. Αυτό είναι το ανώτατο που μπορεί να κάνει ο ΔΟΕ. Ε, βέβαια είναι ένα βήμα που δεν έγινε με μεγάλη ευκολία γιατί τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν εις βάρος του Κατάρ. Όμως ε, ε, εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες διαλόγου ως ε, ΔΟΕ και κυρίως μετά την κατάρρευση του Πλάζα δεν διαπιστώσαμε να υπάρχει κάποια σοβαρή προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα κράτη-μέλη να στηρίξουν αυτήν την ε, έρευνα του ΔΟΕ. Και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει και αυτή η έρευνα GSP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και τελειώσατε και στην ώρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο τον κύριο Μπούχαρτ που ε, αντικαθιστά τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, ε, πρέπει να σας πω ότι οι αριθμοί που ακούσαμε σήμερα μας εντυπωσίασαν, γιατί ακούσαμε ότι έγινε λόγος ε, για εξοικονόμηση 2 δισεκατομμυρίων, αύξηση του 6% και το Μπαγκλαντές ε, το 2024 πλέον δεν θα χαρακτηρίζεται ως ε, least developed country. Ε, δηλαδή με βάση τους αριθμούς βλέπουμε μια θετική εξέλιξη. Φαίνεται ότι το GSP σε αυτή την περίπτωση βαντίζει βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν δούμε όμω τον σχετικό κανονισμό GSP θα διαπιστώσουμε ότι δεν πρέπει να περιζόμαστε μόνο στου αριθμού, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε και την ε, ανάπτυξη τη κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται ε, στα εκτιμώντα 3 και 4 του ε, κανονισμού GSP. Μέχρι τώρα όμω πολλά δεν έχουν αναφερθεί. Παραδείγματο χάρη, ακούσαμε για την παραβίαση εργασιακών διατάξεων αλλά κυρίως όσον αφορά θέματα κυβέρνησης και κοινωνίας θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, στον παγκόσμιο ε, χάρτη περί ανοιχτών open doors έχει κατρακυλήσει το Μπαγκλαντές ακόμα πιο κάτω. Το 2017 ε, υπήρχε ε, μια, υπήρξε μια αλλαγή των ε, ε, σχολικών βιβλίων. Πρέπει να μην υπάρχουν χριστιανικά ή Ινδουιστικά ονόματα και το 18 είχαμε ε, ένα δις ε, δωρεά για τζαμιά σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα θρησκευτικά στοιχεία και αν δούμε λιγάκι το τι γίνεται στην κυβέρνηση και εκεί οι εξελίξεις δεν είναι ικανοποιητικέ. Υπάρχουν πολλά επικριτικά που ακούστηκαν σήμερα πέρα από τα οικονομικά. Εν τω μεταξύ το Μπαγκλαντές έχει κατρακυλήσει, αυτά είναι τα στοιχεία του 2018, στη θέση 149 από τις 180 χώρες όπου μετρήθηκε η ε, διαφθορά. Οι κυβερνητικοί φορείς είναι οι ε, πλέον διεφθαρμένοι και ήδη το 2004 συστήθηκε μια επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μέχρι τώρα όμως δεν σημειώθηκε καμία απολύτως πρόοδος. Τουναντίον φαίνεται ότι η αντιπολίτευση στη χώρα όλο και περισσότερο δέχεται πιέσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και τα οποία κατά την άποψή μου μέχρι τώρα δεν ετέθησαν επιτάπητος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και τώρα οι σκιώδεις εισηγητές έχουν το λόγο. Εκ μέρους του ΕΛΚ δεν βλέπω να έχουμε κάποιον σκιώδη συζητητή. Άγνες Γιούργενς εκ μέρους ε, των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους εσάς που πήρατε το λόγο για να μιλήσετε για τον Μπαγκλαντές. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εμπλοκή του με αυτό το διάβημα για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας των Μπαγκλαντές είναι κάτι που χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω, να Είμαι κοινική ή αισιόδοξη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει ελευθερία του συνέρχεσθε. Οι δηλώσεις των εργοδοτών και των συνδικάτων και των σωματείων είναι σαφείς. Παραμένει ένα μπλοκάρισμα στην καταχώρηση των συνδικάτων και οι διζώνες μεταποίησης προϊόντων με αποκλειστικό αντικείμενο της εξαγωγές το μόνο που κάνουν είναι να επεκτείνονται και να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερα εδάφη στο Μπαγκλαντές ενώ τα σώματα επιθεωρητών εργασίας δεν έχουν αναπτύξει τις δυνατότητές τους αν υπάρχουν που και αυτό δεν είναι βέβαιο. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε ζητήσει Για πλήρη έρευνα EPA, για το κατά πόσο οι επίσημες αρχές του Μπαγκλαντές δικαιούνται αυτό το προτιμησιακό καθεστώς της εμπορικής δραστηριότητας με τίτλο «Οτιδήποτε εκτός από όπλα». Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 μας είχε απαντήσει και μας είχε πει τα εξής «Κοιτάξτε, κάνουμε διάλογο με τον Μπαγκλαντές, θα ασκήσουμε πίεση» και ούτω καθεξής. Και αν δω τις δηλώσεις στο τύπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου μήνα, βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία για χρονοδιάγραμμα και υπάρχει και ο δικός χάρτης και ούτω καθεξής. Πόσο αξιόπιστος είναι, πιστεύετε, ο δικός χάρτης και όντως θα μας οδηγήσει στο τέλος αυτής της ασυλίας που υπάρχει στις ε, ζώνες μεταποίησης με προορισμό της εξαγωγές. Υπάρχουν αληθινές ανησυχίες για την ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε, για το EPA. Ενδεχομένως υπάρχουν επιθεωρήσεις αλλά αν οι επιθεωρητές εργασίας δεν είναι εδώ ή δεν, ε, δεν βρίσκονται επί τόπου δηλαδή ή δεν αμείβονται σωστά, πώς θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αυτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επευθύνουμε τώρα στον πρέσβη του Μπαγκλαντές για να το ρωτήσω το εξή Θα πάρετε στα σοβαρά τον οδικό χάρτη και το, και το χρονοδιάγραμμα. Μας έχετε υποσχεθεί, μας έχετε δώσει υποσχέσεις στο παρελθόν. Το παίρνετε στα αλήθεια σοβαρά. Και τελευταίο σχόλιο που έχω να απευθύνω στον πρέσβη του Μπαγκλαντές είναι το εξής. Πώς ετοιμάζεστε για την κατάσταση μετά το 2024 όπου θα βγείτε από τον κατάλογο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών γιατί οι προσδοκίες ε, από την κυβέρνηση μιας τέτοιας χώρας που έχει βγει από αυτόν τον κατάλογο είναι ακόμα υψηλότερε σε σχέση με, ένα, με μια συμφωνία εμπορική που να περιλαμβάνει οτιδήποτε εκτός από τα όπλα. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο εργασιακός κώδικας πράγματι ο εργατικός κώδικας πράγματι βρίσκονται, είναι θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και καλό θα ήταν να μάθουμε περισσότερα από το πρέσβη. Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή νομοθεσία. Θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρθηκε στο κοινό ανακοινωθέ τύπου στην ένατη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής. Στην πρώτη τελευταία παράγραφο αναφέρεται ότι η μελλοντική αποχώρηση του Μπαγκλαντές από τον κατάλογο των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών θα μπορούσε να είναι υποφελής για τα πιο ευπαθή τμήματα της κοινωνίας. Καλό ακούγεται, αλλά τι σημαίνει ακριβώς ποιο, σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα βγει το Μπαγκλαντές από αυτό το κατάλογο, πώς αξιολογείται και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα πιο ευπαθή ή όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όπως αναφέρει το ανακοινωθέν, θα ωφεληθούν πράγματι από αυτόν τον αποχαρακτηρισμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα από τους Πράσινους. Πράγματι, για αυτό το σύμφωνο ήταν πολύ ψηλέ οι προσδοκίες. Θυμάμαι ένα βράδυ στην Ολομέλεια συζητούσαμε το θέμα με την Επίτροπο Μάλστρομ, θα το θυμάστε και εσείς Πρόεδρε, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από μία από ε, τέτοιε συσκέψει και συνεδριάσεις και δεν, είχε, δεν εμφορεί το καθόλου από εορταστικό κλίμα. Η εντύπωσή μου είναι ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές θα πρέπει να ακούσει τη βιομηχανία πολύ προσεκτικά Ευχαριστώ το, το, σύνδεσμο για το εξωτερικό εμπόριο και τον εκπρόσωπο ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι πράγματι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτές τις μετερρυθμίσεις και μάλιστα πολύ σοβαρά, να το πάρει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα για τον, για τον εργατικό κώδικα και την ελευθερία του ε, συνέρχεστε. Και είναι θαυμάσιο το ότι το λέτε εσείς αυτό. Και είναι θαυμάσιο το ότι λέτε αν ανοίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάκελο ερευνητικό θα στηρίξετε τα συμπεράσματα. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Ακούσαμε τα ωφέλη και μάθαμε ότι η επόμενη συνάντηση στο Compact θα είναι το 2020. Ακούσαμε ότι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περιμένει, να είναι πιο αποτελεσματική από τις προηγούμενες. Θα πρότεινα λοιπόν να υιοθετήσουμε ψήφισμα ή να υποβάλουμε ε, ερώτημα επίσημο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για αυτό το θέμα. Το εκτιμούμε το Compact πάρα πολύ. Έχουμε καλέσει την Επιτροπή επανειλημμένως να το υιοθετήσει σαν μέθοδο και στις σχέσεις της με άλλες χώρες. Ε, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στο Αμφόρης, ε, αυτό το σύνδεσμο για το εξωτερικό εμπόριο ασχολείστε ε, ε, με το να επεκταθεί στον τομέα της ενδυμασίας και της κλωστοεφαντουργίας η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια. Ασχολείστε αυτή τη, με αυτή τη συζήτηση, συμβάλλετε. Εσείς παρακαλώ, δεν έχω κάτι να προσθέσω κύριε Πρόεδρε. Και τώρα η κυρία Σαβατσίνη. Εν συντομία. Και εγώ θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Για το Σύμφωνο Αηφορίας και Βιωσιμότητας, δεν έχουμε πρόσφατα στοιχεία για την ετήσια αξιολόγηση. Συνεχίζει να γίνεται ετήσια αξιολόγηση και πότε προγραμματίζεται. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση στον πρέσβη. Παρόλο που έγιναν βελτιώσεις στα πρότυπα στο Παγκλαντές, μειώνονται οι τιμές. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί αν μια χώρα υποτίθεται συνεχίζει να προσπαθεί, παρόλο που παραμένουν τα πολλά τα προβλήματα, ε, συνεχίζει να προσπαθεί ε, να αυξήσει τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας, τότε γιατί συνεχίζουν να μειώνονται οι τιμές των ρούχων. θα πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσει των Μπαγκλαντέ να αμείβονται με τη σωστή τιμή για το προϊόν τη εργασία τους. Ευχαριστώ κύριος Χέλμουντ Σόλτς. Και εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση η οποία εκτελήσεται στην κοινωνία του Μπαγκλαντές εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη γενοκτονία που συνέβη τον περασμένο αιώνα στη χώρα αυτή και στη συνεχιζόμενη προσπάθεια να αφυπνιστεί η νέα γενιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες και μέσα από το Μουσείο για την Απελευθέρωση. Πώς αυτό δεν αντιφάσκει με το υφιστάμενο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα για το, τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα κάθε πολίτη στη χώρα αυτή. δεν θα έπρεπε να αλλάξει η, η συζήτηση στην κοινωνία. Συζητήσαμε τους εκπροσώπους του Ανφόρη και τους εκπροσώπους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ως Κοινοβούλιο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις μη ικανοποιητικές εξελίξεις ε, έξι χρόνια μετά την, το συμβάν στο Random Plaza, για να ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω την ερώτηση της Αγνής. Όλοι ξέρετε ότι είμαι ε, Γερμανός και από την περιοχή από την οποία κατάγομαι εφημιζόμαστε για την υπομονή μας. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε όσο να τον πιο ρεαλιστές Έξι χρόνια μετά όμως. Έξι χρόνια διαπραγματεύσεις. Για κατάταξη, για χαρακτηρισμό, για βαθμολόγηση και ούτω καθεξής. Ε, τίποτα δεν συμβαίνει. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στις με, ζώνες μεταποίησης με προορισμό με αντικείμενο της εξακογές. Στον οδικό χάρτη ποια είναι τα βασικά στάδια, τα σημεία καμπής, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες δράσεις εάν δεν περαστεί το εκάστοτε στάδιο και αν δεν σημειωθεί η αντίστοιχη αναμενόμενη και προσδοκόμενη πρόοδος. Αυτό είναι και το καθήκον του εις μυστηριώδους θέσης του Chief Trade Law Enforcement Officer που θα δημιουργήσετε. Σιγά σιγά χάνουμε την υπομονή μας, ξέρετε. Και όλα αυτά τα απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρέφομαι τώρα στον πρέσβη του Μπαγκλαντές. Θα έχετε ε, GSP ε, Plus μετά το 2024. Δέχεστε και έρευνα με βάση το EPA. Ο Νίκος πρώτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη για τα ερωτήματά τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο πιο βασικό ερώτημα. Ποια είναι η αξιοπιστία του οδικού χάρτη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Και πολύ καλά κάνετε και μου το ρωτάτε αυτό. τη διαδικασία του EBA δεν την ξεκίνησαν πριν από 26 χρόνια, αλλά το 2017 και πιστεύω ότι φτάνουμε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Έχουμε στείλει πολύ ισχυρά μηνύματα όταν ήμασταν στην ΤΑΚΑ για το ότι επήγει η ανάληψη άμεσης δράσης. Ελπίζουμε ότι αυτός ο δικός χάρτης μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πρώτον, διότι θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και ειδικών. Έχουμε καταστήσει σαφές το γεγονός ότι δεν θα περιμένουμε την πλευρά του Μπαγκλατές να μας παρουσιάζει αλλαγές και να μας λέει ότι έχουμε κάνει αλλαγές αλλά δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτό δεν μας φτάνει πια να είμαστε δηλαδή παθητικοί δέκτες. Οι, δικοί μας εργαζόμενοι και τα για θέματα απασχόλησης θα εμπλακούν στην σύνταξη του οδικού χάρτη. Αυτό καταρχάς. Και δεύτερον, ε, στείλαμε ηχηρό μήνυμα για τα χρονοδιαγράμματα είπαμε ότι ε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα 12 έως 18 μήνες. Είναι επίγουσες δράσεις αυτές που πρέπει να αναλυφθούν. Αυτά έχουμε υπόψη μας. Οι εμπειρογνώμονε και οι δικοί θα συνεδριάσουν, θα συναντηθούν και θα συντάξουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Και αν χρειάζονται περισσότερα τεχνικά στοιχεία, ευχαρίστω θα στραφώ στους αρμόδιους συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση για να σας τα δώσουν. Για το ερώτημα τώρα ε, για τον αποχαρακτηρισμό του Μπαγκλαντές από την κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, Πράγματι, αν οι Ηνωμένε Πολιτείε λάβουν μια τέτοια απόφαση, και αν αυτή η απόφαση ισχύσει το 2024, υπάρχει μεταβατική περίοδος βάσει του GSP Plus τριών ετών, άρα το 2027 ε, το Μπαγκλαντές δεν θα έχει πια το πρωτομησιακό EBA, αλλά θα έχει το απλό GSP ε, γενικευμένων ε, προτιμήσεων και μικρή μείωση των δασμών MFN. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό, ε, ακούσαμε την απάντηση των αρχών, ακούσαμε και τον πρέσβη σήμερα σήμερα δεν, δεν πληρούν τα κριτήρια διαθεσιμότητας και είπαμε ότι ο καλύτερος νίγορος ε, υπεράσπισης της υπόθεσης τους γιατί θα πρέπει να πιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις EPA για να προχωρήσουμε ένα πρόγραμμα πολύ πιο αυστηρό, γιατί το GSP Plus καλύπτει πάρα πολλά πράγματα και τη διαφθορά, για παράδειγμα. Άρα, εμείς του στείλαμε το εξής μήνυμα, ξεφορτωθείτε τα όλα αυτά, τελειώνετε για να πείσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το ότι φιλοδοξείτε να μπείτε στο ε, GSP Plus. Τώρα για το reporting Πότε θα γίνει η επόμενη αξιολόγηση για το EBA. Έκθεση θα δημοσιεύσουμε τον Ιανουάριο του 2020, σε λίγους μήνες. Κάθε δύο χρόνια το κάνουμε για τις χώρες GSP+. Για πρώτη φορά θα συμπεριλάβουμε και κεφάλαιο για τις χώρες EBA. Πιο λεπτομερή περιγραφή των ενισχυμένων δεσμεύσεων με τις τρεις αυτές χώρες, Μπαγκλαντές, Καμπότζη και Μιανμάρ. Και θα τα δημοσιεύσουμε βέβαια αυτά. Τώρα για το σύμφωνο για την αηφορία θα το αξιολογήσουμε πριν την επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο ή Μάιο του 2020. Ευχαριστώ. Απρέσβη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από πού να ξεκινήσω τόσες πολλές ερωτήσεις και τόσα πολλά αιτήματα προς διευκρίνηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το Μπαγκλαντές επανειλημμένο στο παρελθόν έχει αποδείξει πως λαμβάνουμε σοβαρά τις δεσμεύσεις μας. Και εκείνο από αυτό. Πρόσφατα είχαμε την κοινή επιτροπή και συμφωνήσαμε ότι θα συνεργαστούμε για να βρούμε κοινέ λύσεις στα εκρεμή προβλήματα. Μαζί με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό. επίσης, το Μπαγκλαντές, αντιλαμβάνεται ότι έχουμε σχέσεις φιλίας με την Ένωση. Δεν είναι μόνο το EBA, το Everything But Arms. Και αυτό είναι σημαντικό για εμάς και όλα αυτά τα κρατάμε στο μυαλό μας. Έχουμε όμως και ένα καλό ιστορικό επιδόσεων, δηλαδή έχουμε τηρήσει και σεβαστεί όλες μας τις δεσμεύσεις. Άρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως το Μπαγκλαντές θα συνεχίσει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Νιούμαν. Ευχαριστώ. Για να διευκρινίσω κάτι, ε, επειδή κυρία Χάουταλα έθεσε ένα ερώτημα αναφερόμενη στις διάφορες πρωτοβουλίες των κρατών μελών για τη δέωση επιμέλεια σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό ήταν, κύριε Χάουταλ. Ναι, και αυτό, αλλά και τη συνεχιζόμενη και θα έλεγα όλο και πιο έντονη συζήτηση αυτών των ε, εμβαλωματικών νομοθετημάτων Γερμανίας, Ελβετίας, Φιλανδίας, ε, Αντί αυτών να έχουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο σε επίπεδο ένωση Η τι πρεσβεύει. Απάντηση. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο σε ό,τι αφορά τη δέωση επιμέλεια για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα είναι και στην επόμενη θητεία βασικό στόχο. Είναι και στο θεματολόγιο του 2024, στο οποίο, ε, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Πράγματι, καλό είναι να υπάρχει ε, μια ενιαία, οναρμονισμένη ε, προσέγγιση. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την Βαλεντίνα Μπολονιέζε, τη συνάδελφό μου κυρία Χάουτα, λέγε προς τις λεπτομέρειες. Ωραία, μάλιστα. Ακούστε, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θέλουμε την ενωσιακή αυτή προσέγγιση και παραμένουμε σε επαφή για τα λοιπά. Κυρία Σαχάν. Δεν έχω άλλα σχόλια πέραν του ότι θα μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό τον οδικό χάρτη πέραν των δεσμεύσεων όμω, πρέπει να βλέπουμε και αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα τα αιτήματα, σε αυτή τη φάση τα έχουμε ακούσει, έχουν διατυπωθεί επανειλημμένω. Άρα η δέσμευση, η προσήλωση ε, δεν αρκεί να λέγεται ότι υπάρχει, πρέπει να αποδεικνύεται με έργα, με πράξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Πρέσβη, ναι, βεβαίως υπάρχει φιλία, υπάρχει σχέση φιλίας, ε, πραγματικά σοβαρή και ριζωμένη σχέση φιλίας. Αλλά ακριβώς μεταξύ φίλων πρέπει να αναφέρονται με ανοιχτό ειλικρινή τρόπο και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και έτσι θα συνεχίσουμε με αυτή την ανοιχτή συζήτηση για να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε. Και σίγουρα οι υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν για το EBA ε και ελπίζω και στο πλαίσιο μελλοντικά του GSP+. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημείο 25, 24, λέει ο και προχωρούμε στο 25. Uh, λοιπόν, ο κύριος Κλάρκ ε, ε, δεν είναι εδώ. Ε, θα έρθει σε πέντε λεπτά. Και παρότι δεν το συνηθίζω να κάνουμε διάλειμμα, κατ' εξαίρεση θα κάνουμε διάλειμμα πέντε λεπτών. Αλλά αυστηρά πέντε λεπτά παρακαλώ. So, dear members, please take your seats. Καθίστε παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. And Mr. Clark has arrived and he is also now on his... Ήρθε ο κύριος Κλάρκ. Να τον καλωσορίσουμε. Clark, Από πού μας έρχεται? Από την Κίνα. Ήρθε απευθεία από το αεροδρόμιο. Ήταν στην Κίνα όπου και συνήφθη συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ένα θέμα που είναι για καιρό στην ε, ημερήσια διάταξη. Και θυμάμαι όταν είχαμε στείλει μια αποστολή τη Επιτροπής μας στην Κίνα και το είχαμε συζητήσει με τις κινέζικες αρχές το θέμα. Και στην τελευταία διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα ε, ανελήφθησαν κάποιε δεσμεύσει και επιτέλου τώρα έχουμε συμφωνία επιτάπητο που στα σημείο, στο σημείο που έχω εδώ λέει ότι αποτελεί σταθμό αυτό στις οικονομικές σχέσεις. Είναι έτσι Τζον ή όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα έφτανα στο σημείο να τη χαρακτηρίσω σταθμό, αλλά μια πολύ θετική εξέλιξη σίγουρα είναι στις σχέσεις μας με την Κίνα. Είναι η πρώτη διεθνή εμπορική συμφωνία με την Κίνα και αυτό έχει τη σημασία του, πέραν του περιεχομένου της συμφωνίας αυτό αυτό. Η Επιτροπή σας γνωρίζει τις διάφορες ε, μορφές ε, του κειμένου. Στην Κίνα τη Δευτέρα καταλήξαμε και ο Επιτρόπος Χόγκαν και ο Κινέζος ομόλογος ε, προέβησαν σε δημόσια δήλωση την Τετάρτη στο Πεκίνο και σήμερα τα μέσα βρίθουν δημοσιευμάτων η Κίνα είναι πολύ σημαντική αγορά για τις ε, γεωγροδιατροφικές μας εξαγωγές. Δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, 14 δις ευρώ εξαγωγών το χρόνο και αυξάνεται αυτό το νούμερο. Με αυτή τη συμφωνία θα έχουμε υψηλού επίπεδου προστασία και κάτι πολύ σημαντικό, προστασία των εικονικών ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων σε τρόφιμα και ποτά οι Κινέζοι καταναλωτές ε, όλο και περισσότερο εκτιμούν ε, την αυθεντικότητα και την ποιότητα των ευρωπαϊκών ποτών και τροφίμων και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει να εξάγουμε περισσότερο και να ε, παρέχουμε ευρωπαϊκά προϊόντα στους Κινέζους καταναλωτές. Θα βοηθήσει ιδίως στους ευρωπαϊκούς τους ευρωπαίους παραγωγούς ε, τροφίμων και τους αγρότες μας. Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με τελευταία φορά που το συζητήσαμε. Η πρώτη φάση προβλέπει προστασία 100 ονομασιών και γραφικών ενδείξεων. Τα πιο γνωστά από εμπορική και πολιτική σημασία είναι και ε, εκατοστή αντίστοιχα ε, προϊόντα κινέζικα. Πολύ ε, νόστιμα προϊόντα από την Κίνα θα προστατεύονται και αυτά πλέον. Έχουμε τη συμφωνία TRIPS και το άρθρο 23. Σε αυτό το επίπεδο θα είναι η προστασία, πολύ υψηλό επίπεδο, για να μην υπάρχουν παραπλανητικές ενδείξεις για τον καταναλωτέ. Έχουμε τη δυνατότητα συνύπαρξης γεωγραφικών ενδείξεων με εμπορικά σύμπτωτα που ήδη υπάρχουν, με σήματα κατατεθέντα δηλαδή, και σε μια δεύτερη φάση τη συμφωνίας, τέσσερα χρόνια μετά τη θέση ισχύ, 175 ονομασίες ε, ενθεν θα μπουν ε, και αυτές αυτοκαθιστώς προστασίας. Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόπτικη, 275 δηλαδή προϊόντα, 275 ονομασίες από την Κίνα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η συμφωνία. Προσπαθούμε στο δυνατόν πιο γρήγορα να προχωρήσουμε σε στο επίπεδο του Συμβουλίου, ώστε το 2020 και στις αρχές κιόλας του έτους ε, να επιληφθεί το Κοινοβούλιο. Η κινέζικη πλευρά έκανε πολύ θετική ε, παρουσίαση της απόφασης, της συμφωνίας αυτής, ε, την παρουσίαση δηλαδή ως κάτι πολύ θετικό, ότι θα προστατευτούν έτσι τα ποιοτικά του τρόφιμα, ε, θα προστατευτούν και τα ευρωπαϊκά πνευματικά δικαιώματα και θεωρούν ότι αυτό ανοίγει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας πολύ σημαντική συνθήκη, πιο σημαντική των τελευταίων ετών. Και συμφωνούμε σε αυτό και εμείς νομίζω ότι ε, αυτή η καμπή, αυτή η νέα τροπή στις σχέσεις ε, θα ε, είναι ίσως πράγκελος και άλλων συμφωνιών, όπως παραδείγματος χάρη επενδυτική συμφωνίας με την Κίνα. Άρα και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς γεωπολιτικής σημασίας αυτή η συμφωνία έχει ε, τη σημασία της, έχει την αξία της και ελπίζω οι ευρωβουλευτές ε, να βρουν κάτι που να τους ε, ικανοποιεί και να τους προκαλεί το ενδιαφέρον από αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και που ήρθατε μάλιστα κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Κύριε Βίνκλερ, είστε ικανοποιημένο. Πρόεδρε, έμεσα ναι, αλλά ε, πραγματικά δεν είναι τυχαίο που και εγώ αναφέρω στι δικέ μου σημειώσει ότι πρόκειται για μια συμφωνία ορόσημο. Φαίνεται ότι ανάμεσα στου σοσιαλδημοκράτε και το ΕΛΚ υπάρχει τελικά συμφωνία τουλάχιστον από αυτού του θέματο. Νομίζω ότι αυτά που μόλι ε, τώρα ακούσαμε από το Διευθυντή τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ σωστά ότι πρόκειται για μια νέα φάση στη σχεση Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Ελπίζω αυτό να επαληφθεί ε, και θέλω να ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία περί γεωγραφικών ενδείξεων ε, θα βελτιώσει τις εμπορικές μας σχέσεις. Ε, έχουμε μηνύματα, τα πήραμε αυτή την εβδομάδα από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Κογκρέσου της Κίνας, ο πρόεδρος Ιτζιπίν. Νομίζω ότι και αυτός δεν δεσμεύτηκε ακριβώς, αλλά έκανε κάποιες πολιτικές δηλώσεις για το ότι το 2020 είναι δυνατόν να υπάρξει μια διμερή συμφωνία επενδύσεων. Δεν είναι ακόμα δέσμευση, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία περί γεωγραφικών ενδείξεων που υπογράφτηκε αυτή την εβδομάδα στην Κίνα ήταν το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ε, θα περάσει μια νέα φάση ε, και αυτές οι πάνω από 100 ενδείξεις θα συμπληρωθούν, θα γίνουν ακόμα περισσότερες, άρα δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εγώ θα πρότεινα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να μας ενημερώνει, βεβαίως και το πράττει αυτό η Επιτροπή, ε, διότι ίσως ε, και εμείς να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια επιτυχημένη ιστορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επελώς περιοχές όπου οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Γεωργίας, ο οποίος σε λίγες μόνο εβδομάδες θα είναι βέβαια ε, Επίτροπος Εμπορίου. Και αυτή είναι μια πολύ καλή μετάβαση για τον κύριο Χόγκαν. Από τα γεωργικά θα περάσει στα εμπορικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους σκιώδεις εισηγητές. Εκ των Σοσιαλδημοκρατών, η ε, κυρία Πενιέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον πρόσωπο, τον, κύριο Κλάρκ και τον κύριο Βουίνκλερ. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να ε, εκφράσουμε τις ευχαριστήσεις μας προς ε, τον κύριο Χόγκεν για την ομάδα του. Ή πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι πράγματι σήμερα. Το θέμα είναι το ποιοτικό στοιχείο πιο πολύ, το ποσοτικό, γιατί ανοίγει δρόμους και θα υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη αξιοπιστία, αναγνώριση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό συνδέεται και με τον τρόπο ζωής μας, και με την ε, υπεράσπιση της ε, αγροτικής οικονομίας ε, και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Συμφωνώ λοιπόν και εγώ ότι αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή τη συμφωνία. Το σημαντικό είναι τώρα να δούμε ότι αυτή η μεταβατική περίοδος για τα 175 χρόνια θα πρέπει νομίζω να επεκταθεί πέραν των 4 ετών για να περιληφθεί και άλλα προϊόντα, χωρίς που δεν είναι ακόμα μέλη ε, της Ένωσης ή ε, κράτη τα οποία ήταν τότε όταν διαπραγματεύτηκε η κρατη τα μέλη. Νομίζω ότι προβλέπεται μία αναθεώρηση αν προκύψουν συνθήκες που ε, θα καταστούν πάρει την προστασία άλλων γεωγραφικών ενδείξεων. Αν δηλαδή υπάρξει πρόβλημα ότι μπορεί να αντιγράφονται, να είναι αντικείμενα απομίμησης και τα λοιπά, κάποια προϊόντα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Αυτή η αναθεώρηση πώς προβλέπεται να γίνει και όπως πάντα ε, με τις εμπορικές συμφωνίες. Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της εφαρμογής, της υλοποίησης. Ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί που θα σας επιτρέψουν να εγγυάστε ότι τα προϊόντα που θα τη χάνουν προστασία ό,τι αφορά τη γραφική τους ένδειξη, δεν θα μπορεί εύκολα να παραποιούνται, να γίνονται απομιμήσεις αυτών δηλαδή. Τι προβλέπει η συμφωνία και πώς οι εφαρμογές της μπορεί να, να ελεγχθεί σε αυτό το σημείο. Σίγουρα ελπίζουμε να έχουμε και την επενδυτική συμφωνία. Έτσι ξεκινάει ένα νέο πλαίσιο όπου η Κίνα θα σέβεται τους κανόνες διεθνούς εμπόριου και θα μας βοηθά και μας να βγούμε από το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα ο ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Κάριν Κάλσμπρο από τη Ρωμάδα Ρινιού. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Βεντράν ε, ζητά συγγνώμη, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα στη συνεδρίαση και έπρεπε να επιστρέψει στην εκλογική της περιφέρεια. Είχε ηλυμένες υποχρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ να αναφέρω κάποια θέματα που θα ήθελα να θίξει η ίδια. Ε, η ολοκλήρωση αυτής της ε, διμερού ε, συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη γιατί αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η τεχνογνωσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους καλλιεργητέ, τους αγρότες, να προστατεύσουμε ε, θέσει απασχόληση. Εμβαθύνονται οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στι διαπραγματεύσει με την Κίνα, να ακολουθήσουμε το το πνεύμα της αμοιβαιότητας, ε, της ε, πολυμέρειας, ε, να προσπαθούμε να εντάξουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Η Συμφωνία που ολοκληρώθηκε χτες δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί το εμπόριο, να δημιουργηθούν νέα ωφέλη, να υπάρχει πλήρης προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων. Προσβλέπουμε στο να ξεκινήσει η μελέτη σχετικά με τη Συμφωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση ε, σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ε, για να ε, βρούμε την, να καταλήξουμε σε δέσμευση και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε να λυθούν τα θέματα που υπήρχαν κατά το παρελθόν σε αυτή την τόσο επίμαχη ζώνη. Ε, πράγματι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λυθούν ε, τα διάφορα θέματα. Ε, εγώ νομίζω ότι ήδη έχουμε συγκεκριμένες εξελίξεις για το πώς ακριβώς θα εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή σε μια χώρα όπως είναι η Κίνα, σε όλες τις, τις επαρχίες και περιφέρειες. Εκεί τα πράγματα ποικίλουν, είναι διαφορετικά, δεν είναι παντού τα ίδια. Και το δεύτερο που θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα κινέζικα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν και πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να καταναλώνουν κάποια ειδικά κινέζικα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Λέει η κυρία Αγγιλέρα Γκαρθία. Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια. Πολύ σωστά τα είπε. Θέλω να εκφράσω κάποιες εκτιμήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Γεωργίας, η οποία στη συνέχεια θα κληθεί να συντάξει γνωμοδότηση με βάση τις ε, κείμενες διαδικασίες. Να τονίσω κάτι που για μας είναι σημαντικό. Έχουμε περάσει από μια κατάσταση κατά την οποία υπογράφονταν συμφωνίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις. Από αυτή την κατάσταση τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση πολύ πρωτοποριακή μπροστά από την νομοθεσία μας. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια χώρα με την εξαιρετική μας νομοθεσία και είναι ε, ε, μια κίνηση αυτή, ε, μια έναρξη για να διαμορφωθούν οι μελλοντικέ εμπορικές μας σχέσεις με μια χώρα που μας ενδιαφέρει, όπως είναι η Κίνα. Θεωρούμε δηλαδή εμείς ότι έχει γίνει ένα βήμα μπροστά, σημαντικό, με τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις σε αυτή τη συμφωνία. Για μας είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Η Γενική Διευθύνση Γεωργίας έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι μια δουλειά πολλών ετών και θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες. Το σημαντικό για εμάς, όχι μόνο για την κινέζικη αγορά που είναι πολύ μεγάλη, αλλά το σημαντικό για εμάς είναι να προστατεύσουμε και τις μελλοντικέ γεωγραφικές ενδείξεις, 175 τώρα και 275 στη συνέχεια. Θα είναι ένα προηγούμενο πολύ σημαντικό και για την αγορά των ΗΠΑ και για την αγορά της Λατινικής Αμερικής, όπου υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις σε σχέση με κάποιες από τις σημαντικές μας ονομασίες προέλευσης. Είναι πολύ θετική δηλαδή αυτή η εξέλιξη, όχι μόνο για το κινέζικο πλαίσιο, αλλά γιατί μας αναγνώρισε ε, την γεωγραφική ένδειξη ποιότητας ε, που θα μπορούμε να επικαλαστούμε και με άλλους εταίρους και σε άλλες αγορές που μας τις αμφισβητούν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι. Έγινε τεράστια προσπάθεια και θεωρούμε ότι αυτός ο τρόπος σύναψης νέων, ε, νέος τρόπος σύναψης ε, εμπορικών συμφωνιών είναι πρωτοποριακός από πλευράς νομοπαρασκευαστικής και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Νικολά Ντάντι παρακαλώ. Ο Νίκολα, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να πω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με αυτή τη συμφωνία. Όχι μόνο ε, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι ε, κατά τα επόμενα έτη θα προσθεθούν και άλλες ενδείξεις και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο κυρίως για το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία με μια χώρα ε, μία συμφωνία η οποία αφορά σε αυτή τη φάση την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό είναι σημαντικό ότι το κάνουμε με την Κίνα. Το έχουμε κάνει βέβαια ε, και σε άλλες περιπτώσεις ε, και πρέπει να υπάρξουν και άλλες συμφωνίες με την Κίνα γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας αλλά ε, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και ε, συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικό το ότι και εμείς αναγνωρίζουμε βέβαια κάποιες ε, κινέζικες γεωγραφικές ενδείξεις ε, και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε και αποδεικνύουμε ότι σκεπτόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός. Από τις ε, 31 γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες προστατεύονται στην Ευρώπη. Ε, περίπου οι μισές είναι αγροδιατροφικές, άλλες δεν είναι ε, αγροτικές. Κάπως πρέπει να το σκεφτούμε βέβαια αυτό. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το δικαίωμα ε, να, με βάση τη συνθήκη της Γενέβης και τη Συμφωνία της Λισαβόνας σχετικά με την ονομασία ε, και τις προελεύσεις ε, και τις, ε, τις συμφωνίες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε το δικαίωμα λοιπόν να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τη δική μας την νομοθεσία για να αποδειχθεί ότι και η Ευρώπη στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων ενδιαφέρεται και για άλλα προϊόντα και όχι μόνο για τα αγροδιατροφικά. Το Κοινοβούλιο νομίζω με 650 ψήφους ε, ψήφισε υπέρ σε ένα ψήφισμα όπου καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει μία διαδικασία προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να προσθεθεί, να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τις σχέσεις με την ε, Κίνα. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες ερωτήσεις στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θέλω να καταλάβω πρώτον τι είδου προστασία διαπραγματευτήκατε, δηλαδή αυτή η προστασία συμπεριλαμβανομένη και την περίφημη επίκληση των ονομάτων. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, σε τι ακριβώ αναφέρεστε όταν μιλάτε για γεωγραφικές ενδείξεις ή μη αγροτικές. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε τι είναι αυτό το μίσο αγροτικό ή μη αγροτικό. Η Τιτσιάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ε, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, γιατί πράγματι αυτό είναι σημαντικό βήμα προς το εμπρό, προς την ε, πλήρη προστασία και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού μας τομέα στην Κίνα. Είναι ευρύτατος ο τομέας, ε, οι απομιμήσεις, οι παραποίησεις, ε, αυτά είναι μάστιγες για τους ε, παραγωγούς μας. Άρα δηλαδή είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και για πολλούς άλλους λόγους ε, όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα. Νομίζω ότι εξάλλου είναι και πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα αυξηθεί ο αριθμό των προϊόντων που θα προστατεύονται σε διάρκεια τεσσάρων ετών, άρα δηλαδή θα προσταθούν και πολλές ε, άλλες ενδείξεις. Κατά τα άλλα βεβαίως και έχουμε ανησυχίες όπως τις εξέφρασαν ε, και κάποιοι συνάδελφοι γιατί υπάρχουν και προϊόντα που δεν είναι γεωργικά και αυτά θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή γιατί ο ε, διατροφικός τομέας ε, Βεβαίω και είναι σημαντικό, αλλά ίσω όχι και τόσο σε σχέση με άλλα προϊόντα. Ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε, πάντω είμαστε στο σωστό δρόμο. Θέλω να κάνω μία ερώτηση σε σχέση με την περίοδο τη συνύπαρξη. Η παραγωγή είναι λιγάκι ανήσυχη, ε, δηλαδή η περίοδο συνύπαρξη ε, με προϊόντα που θα έρχονται από τι ΗΠΑ και από τη Νέα Ζηλανδία, κυρίω όσον αφορά τα ε, προϊόντα στον τομέα των τυριών και των γαλακτοκομικών κομικών. Ανησυχούμε λιγάκι αυτή την περίοδο, ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε. Συνάδελφοι, βλέπετε αυτό το πορτοκάλι. Έρχεται από μακριά, από άλλη ήπειρο, αλλά ε, σε κάποια μέρη του κόσμου πωλείται ως πορτοκάλι της Σικελίας. Και αυτό δεν είναι σωστό. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με το ε, βίνο μαρσάλα με πάρα πολλά ζυμαρικά τα οποία αποκαλούνται Ιταλικά παρότι δεν είναι Ιταλικά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ποιοτικά προϊόντα της Ιταλίας τα οποία ε, παραποιούνται και αυτά αφαιρούν πόρους από τις επιχειρήσεις μας. Άρα δηλαδή καλό είναι αυτό που υπήρξε αυτή η πρώτη συμφωνία αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο η προστασία να επεκταθεί και σε πολλά άλλα προϊόντα, σε προϊόντα της Νότιας Ιταλίας ε, και των νησιών, ε, γιατί εκεί θεωρώ ότι η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει ε, την ανάπτυξη και θέλω να είμαι σίγουρος ότι αυτά τα πορτοκάλια που θα πουλούνται στο μέλλον ως πορτοκάλια της Σικελίας να είναι πράγματι πορτοκάλια που έρχονται από τη Σικελία και είναι Σικελιανά. Πρόεδρε, προφανώς έγινε ένα βήμα προς τα εμπρός. Εμείς αυτό το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και είναι επίσης και σαφές ότι ορισμένοι που προηγήθηκαν για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων είπαν ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα αγροδιατροφικά, ε, θα πρέπει να προσθεθούν και άλλα προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Όσον αφορά τώρα το σχέση στο σύνολό τους με την Κίνα, Ίσως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευνοϊκή στιγμή ε, για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των απομιμήσεων και των παραποίησεων. Εκεί η Κίνα είναι πρώτη ε, όσον αφορά τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη. Ε, μιλάμε κυρίως για προϊόντα μεταποιημένα. Εκεί δεν υπάρχει διαφάνεια τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο καταναλωτής ε, πρέπει να αγωνιστεί για να καταλάβει ε, από πού προέρχονται όλα αυτά τα προϊόντα που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι σαφές, δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει την προέλευσή τους. Εμείς ε, λοιπόν ως Επιτροπή Διεθνούς Συμπορίου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά περισσότερα και να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς γιατί πρέπει τα προϊόντα να είναι σαφώς από πού προέρχονται ε, και να προστατεύονται από τέτοιου είδους ε, συμφωνίες. Η κυρία Γκιόριχ. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία. και πότε θα δώσει την απαραίτητη συνέχεια το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω να σας θέσω, Τζον, ένα πολιτικό ερώτημα ως Πρόεδρος. Ποια είναι η αποψή σας. Πιστεύετε ότι η Κίνα στρέφεται τώρα περισσότερο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα εκπρόσωπο τη κυβέρνηση μα είπε ότι δεν είναι θέμα το περιεχόμενο τη συμφωνία των Γεωγραφικών Ενδείξεων όταν τη συζητήσαμε, είναι περισσότερο θέμα ροπή τάση. Πρέπει να υιοθετήσουμε την αμερικανική νοοτροπία που μισεί τι γεωγραφικέ ενδείξει. Ή πρέπει να πάμε να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Άγου, α λαμβάνοντα υπόψη ότι έτσι κλιμακόνεται ίσω η ένταση με τι ΗΠΑ. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκομίσει, Τζον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το γεγονός ότι πράγματι αντιστάθηκε στην μεγάλη πίεση από τη ΣΥΠΑ η Κίνα και αποφάσισε να προστατεύσει τις ονομασίες ε, γεωγραφικής ένδειξης διότι καταλαβαίνει ότι δεν θα ήταν σόφρον να ακολουθήσει ε, την αμερικανική άποψη μέχρι τέλους και ότι μπορεί να έχει στην Ευρώπη ε, να βρει ένα σύμμαχο, ένα φίλο και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Συναντήσαμε τον Τζιντζιπίνγκ και τον ε, Υπουργό Εμπορίου χθες σαφέστατα μας είπαν ότι ερμηνεύουν αυτή τη συμφωνία και την αντιλαμβάνονται ως πολύτιμη αυτή καθ' αυτή, αλλά και ως συμβολική ως θεμέλια λίθος αν θέλετε με συμβολική σημασία για περισσότερο επικοδομητικές και θερμές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Άρα υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις που δεν θα πρέπει να παραμελεί κανείς. Εν συντομία να θίξω και δύο-τρία ζητήματα που έθεσαν τα μέλη σας. Ο κύριος Ντάντι έθεσε δύο ερωτήματα. Ποιο είναι το επίπεδο προστασίας της συμφωνίας, απαντώ λέγοντας ότι είναι υψηλό, πολύ υψηλό πάνω από το επίπεδο 23 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και έχουμε και το άρθρο 4 της Συμφωνίας που προστατεύει τις ονομασίες μας σε οποιαδήποτε μέσα και στη συσκευασία και αλλού και στην ετικετοθεσία που ε, προσπαθεί να δείξει ότι ένα αγαθό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης, ο κύριος Ντάντι μας ε, έθεσε ερώτημα για τα ημιαγροτικά. Σε αυτή τη συμφωνία δεν προστατεύουμε μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομική βάση για να το πράξουμε. Θέλω να το καταστήσω αυτό σαφές. Όχι άμεσα, αλλά στη δεύτερη λίστα, στο δεύτερο κατάλογο, προστατεύουμε 14 κινέζικες γεωγραφικές ενδείξεις που εκπορεύονται από ε, γεωργικές πρώτες ύλες. Και αυτό υπάρχει στον αρισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας, παράρτημα 5 της συμφωνίας. Η κυρία Μπέγγεν μου έθεσε κάποια ερωτήματα και απαντώ λέγοντας ότι ως προς την επιφύλαξη που εκφράσατε για τις μεταβατικές περιόδους, για ορισμένα τυροκομικά προϊόντα, η φέτα μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται. Όντως έπρεπε να ε, φτάσουμε σε ένα συμβασμό σε αυτούς τους τρεις τομείς. Πιστεύω όμως ότι το αποτέλεσμα είναι καλό για την Ιταλία και την Ελλάδα. Δηλαδή μετά από έξι χρόνια κανείς στην κινέζικη αγορά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο Ασιάγκο εάν δεν βασίζεται σε Ιταλό ε, ε, παραγωγό. Κανείς δεν μπορεί για τρία χρόνια να χρησιμοποιήσει τον όρο Ρωμάνο ε, άμα δεν μιλάει για πεκορίνο αληθινό. Το αντίστοιχο και για τη φέτα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ε, όλα αυτά με βάση τις μεγάλες πιέσεις που ασκεί ο τυροκομικός και ε, γάλακτοκομικός τομέας από την Αυστραλία, την Νέα Ισλανδία, τις ΗΠΑ, Καναδά. Είναι μια εθνική συνθήκη και πρέπει να περάσει βέβαια από όλη αυτή τη διαδικασία του Συμβουλίου και θα προσπαθήσουμε να ε, να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με το Συμβούλιο μέχρι τα μέσα του 2020. Και Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες και τις κατανοώ απολύτως για την εφαρμογή, για τη θέση σε ισχύ, για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται και υλοποιείται η συμφωνία. Θα έλεγα ότι η Κίνα παίρνει την εφαρμογή της συμφωνίας στα σοβαρά και η εμπειρία που έχω αποκομίσει από τους Κινέζους είναι ότι άπαξ και καταφέρουμε να υπογράψουν κάτι, όντως το παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Έχουν ήδη οργανώσει τη διοίκησή τους έτσι ώστε υπό μία αρχή και υπό μία υπηρεσία να υπάγονται όλα τα διαδικαστικά για το IPR, για τη διανοητική ιδιοκτησία. Η σύμβαση προβλέπει ότι όχι μόνο κατόπιν ετύπηματος του δικαιούχου, αλλά εξοφίτσιο οι κινέζικες αρχές θα υιοθετήσουν κανόνες για να αποσύρουν προϊόντα που δεν περνούν τις προϋποθέσεις από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και έχουμε και τη θέση σε ισχύ των ε, γεωγραφικών ενδείξεων Απόδειξη της καλής τους θέλησης υπ' αυτή την έννοια είναι το εξής. Ως προς τις 175 ονομασίες γεωγραφικής ένδειξης που περιμένουν να ε, τύχουν προστασία στο μέλλον αλλά δεν προστατεύονται αυτή τη στιγμή, έχει αναστείλει η Κίνα ε, το δικαίωμα να υποβάλει κανείς αίτηση να αποκτήσει trademark κατά αυτών των 175 ονομασιών προσωρινά. Ε, και αυτό είναι πολύ θετικό. Σε σχέση με αυτά που λέει η κυρία Ροντρίκε Πινιέιρο, να σας πω ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα δείγμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, αν δεν έχει κανεί εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να φτάσει σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι υψηλό το επίπεδο εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Και πράγματι, όπως είπατε και εσείς, αξιότιμη κυρία Βουλευτής, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει παγκοσμίω ε, το σήμα ποιότητας, την έννοια της ποιότητας και τα υψηλά πρότυπα στα οποία ανταποκρίνονται τα δικά μας ευρωπαϊκά προϊόντα. Και αυτό σε γενικές γραμμές είναι κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο για τα ε, θερμά της σχόλια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριος Βίνκλερ παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Επαναλαμβάνω τις ελπίδες που έχουν εκφραστεί εδώ, ότι δηλαδή το 2020 θα είναι το έτος όπου θα προχωρήσουν πραγματικά οι ευρωκινέζικες σχέσεις. Και πιστεύω ότι η συμφωνία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την ύπαρξη αυτής της ε, συμφωνίας με την Κίνα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το πραγματικά εφικτό. Ευχαριστούμε. This concludes 26 uh, and have a good... Όπερε διδείξε, όπως όλοι οι πολιτικοί και εσείς. Αυτά λοιπόν. 26 ποτά διάφορα. Τίποτα. 27. Επόμενη συνεδρίαση 25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και 2 και 3 Δεκεμβρίου. Καλό μεσημέρι. Καλά να περάσετε μέχρι την επόμενη μας συνεδρίαση.